An alle einen guten Morgen. Jetzt sind so lang... Καλημέρα σε όλου. Νομίζω πω οι περισσότεροι από εσά έχουν έρθει. Στι 12 Νοεμβρίου δημιουργήθηκε η ημερήσια διάταξη. Υπάρχουν αντιρρήσει για αυτή. Όχι. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχουν κάποιες εντρήσεις, τότε νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στα θέματά της. Να σας ενημερώσω καταρχάς ότι σήμερα υπάρχει διερμηνία σε όλες τις γλώσσες, δεν θα τις διαβάσω. Επίσης, η συνεδρία μεταδίδεται ζωντανά από το διαδίκτυο και ελπίζω να έχετε όλοι μαζί σας τις κάρτες ψηφοφορίας διότι θα ξεκινήσουμε με ψηφοφορία. Με θέμα το κλείσιμο των λογαριασμών της ΕΑΣΟ, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για, τον, για το άσυλο. Μπορούμε λοιπόν, μια που λοιπόν ο να περάσουμε απευθείας στην ψηφοφορία. Ψηφίζουμε λοιπόν για το κλείσιμο των λογαριασμών της ΕΑΣΟ. Θα έδινα κανονικά το λόγο στον εισηγητή, αλλά μπορεί να ζητήσει και όποιος άλλος θέλει το λόγο. Εφόσον δεν θέλει καλής, μπορούμε να ψηφίσουμε. Ή όποιος είναι υπέρ, παρακαλώ να το δηλώσει ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 14 ψήφοι υπέρ, 3 κατά, μία αποχή. Πολύ ωραία. Περνάμε στην απαλλαγή για το 2008. Ξεκινάμε με τις κοινέ επιχειρήσεις. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε ένα μέλος του ελεκτικού συνεδρίου μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε, κυρία Γκάλ Πέλτς. Η είναι ο κύριος Μπλουτζίνσκι για τον καθαρό ουρανό. Μετά ο κύριος Λεγκούτκο για το Shift to Rail, την ΣΕΖΑ και τις ε, κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου. Θα δώσω όμως ε, αμέσως το λόγο στην Ιλντίκο. Α, εδώ είστε, εδώ είστε. Έχετε λοιπόν το λόγο και σας ευχαριστώ πολύ προκαταβολικά που θα μείνετε εντό του ορίου των 10 λεπτών. Gibt es noch Schwierigkeiten? Uh, έχετε κάποιο πρόβλημα? Όχι, όχι. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, νομίζω πως όντως υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα με το PowerPoint, την παρουσίαση που είχα ετοιμάσει. Θα ήθελα λοιπόν λίγο χρόνο για να μπορέσω να ξεκινήσω την παρουσίαση. Ωραία, θα ξεκινήσουμε με τους επικεφαλείς των κοινών επιχειρήσεων. Μετά ελπίζω να λυθεί το πρόβλημα. Έχουμε και λέμε... Έχουμε τον κύριο Πίμπουκα από τις Κυψέλες Καυσίμου και Ιδρογόνου, τον Ιωάννη Σφέμα, ο οποίος θα μας παρουσιάσει την δική του κοινή επιχείρηση, ο κύριος Αξελ Κράιμ και μετά θα δώσουμε το λόγο στους δικούς μας εισηγητές, τους κοιόδης εισηγητές και έπειτα θα υπάρχει δυνατότητα να θέσετε ερωτήσεις εφόσον το επιθυμείτε. Ωραία, μπορώ να ξεκινήσω λοιπόν, διότι είναι έτοιμα, έτοιμη παρουσίαση. Ωραία, λοιπόν, χαίρομαι που λύθηκαν τα τεχνικά προβλήματα. Ηλτίκο παλιτσά, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσετε να παρουσιάσω την ετήσια έκθεση για τις κοινέ επιχειρήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018. Για πρώτη φορά υπάρχει μια ενοποιημένη έκθεση για όλες τις κοινέ επιχειρήσεις η οποία έχει χωριστεί σε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει μια γενική εικόνα των κοινών επιχειρήσεων, το κεφάλαιο 2 μετά τα γενικότερα αποτελέσματα των ελέγχων και το κεφάλαιο 3 περιέχει τις ε, δηλώσεις αξιοπιστίας, τις δικές μας γνωμοδοτήσεις και παρατηρήσεις για τις κοινέ επιχειρήσεις. Η έκθεσή μας δημοσιεύθηκε στο, στην ιστοσελίδα του Ελεκτικού Συνεδρίου το Νοέμβριο. όπως προβλέπει το άρθρο 287 της Συνθήκης, έχουμε διεξάγει ελέγχου στους λογαριασμούς όλων των κοινών επιχειρήσεων και ελέγξαμε επίσης την νομιμότητα και την κανονικότητα των συναλλαγών στους λογαριασμούς αυτούς. Σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 του Δημοσιονομικού Κανονισμού, ο έλεγχος της ε, κανονικότητας των λογαριασμών όλων των κοινών επιχειρήσεων υπόκειται, ε, μάλλον θα γίνει από ανεξάρτητους ε, ελεγκτές, εξωτερικούς ελεγκτές. Για κάθε κοινή επιχείρηση έχουμε εξετάσει την ποιότητα των ελέγχων, ιδιαίτερα για τους τομείς που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο. Θα σας πω τώρα δύο λόγια για τις κοινέ επιχειρήσεις. Νομίζω πως όλοι γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται. Οι κοινέ επιχειρήσεις είναι συμπράξεις δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, ε, ομάδων έρευνας και των κρατών μελών. Παίζουν ένα σημαντικό ρόλο ε, σε πολύ σημαντικές ε, πτυχές της ερευνητικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και διασφαλίζουν την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας δημιουργήθηκαν με βάση το άρθρο 187 της συνθήκης και στην περίπτωση της ε, σύνδεξης για την ενέργεια Fusion for Energy της ε, συνθήκης Ευρατόμ. Όπως βλέπετε στη διαφάνεια, το, ο συνολικός προϋπολογισμός για το 2018 ανέρχεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου δηλαδή το 1,5% του συνολικού προπολογισμού της Ένωσης. Οι 7 κοινέ επιχειρήσεις ε, που λειτουργούν υπό τον ορίζοντα 2020 ε, έχουν πλησιασει στην 1.221 ευρώ. Το Fusion for Energy λειτουργεί ε, με βάση τη συνθήκη Ευρατόμ και έχει προπολογισμό 795 εκατομμύρια ευρώ. Οι κοινέ επιχειρήσεις απασχολούν 669 υπαλλήλους και το 2017 676. Η συνολική συνεισφορά της Ένωσης είναι 4 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτό, αυτά αποτελούνται από 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε διάφορες επιχειρησιακές δραστηριότητες εντός ε, του σχέδιου εργασία των κοινών επιχειρήσεων και 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε καθαρές συνεισφορές σε εξωτερικές δραστηριότητες που βρίσκονται όμως εντός του πεδίου εφαρμογή ε, και των στόχων των κοινών επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά του, το βαθμό εφαρμογής ε, των δραστηριοτήτων αυτών βρίσκεται στο 89% του στόχου και ε, κατά το κλείσιμο του προγράμματος και ε, οι στόχοι του ορίζοντα 2020 επίσης δεν έχουν εκπληρωθεί διότι εκεί το ποσοστό εκτέλεσης ήταν 39%. Ας δούμε τώρα με λεπτομέρειες τον έλεγχο. Τι ελέγχθηκε λοιπόν, όπως κάθε χρόνο έγιναν έλεγχοι και έκδοσαμε γνωμοδοτήσεις για την αξιοπιστία των λογαριασμών και την γνωμιμότητα και κανονικότητα των συναλλαγών για το ε, οικονομικό έτος ε, που έληξε στις 31 ε, Δεκεμβρίου του 2018. Πρώτα, αξιοπιστία των λογαριασμών όπως ήδη σας είπα, για όλες ε, τις ε, κοινέ επιχειρήσεις, η αξιοπιστία των λογαριασμών του 2018 ελέγχθηκε από εξωτερικές ε, ελεκτικές εταιρείε. Αξιολογήσαμε την ποιότητα των ελέγχων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και λάβαμε διασφαλίσεις για την ποιότητα της δουλειάς. Αυτά λοιπόν ως προς τον έλεγχο το 2018. Έπειτα νομιμότητα και κανονικότητα των λογαριασμών. Λάβαμε ε, διασφαλίσεις οι οποίες βασίστηκαν ε, σε συστήματα εσωτερικού ελέγχου, τα οποία εξέτασαν ε, τις κύριες διοικητικές και επιχειρησιακές δραστηριότητες. Μετά έγιναν ουσιαστικοί έλεγχοι από δείγματα πληρωμών και άλλων συναλλαγών. Ελέγχθηκε η, εξ, η, ελέγχθηκαν οι εξπόστα ελεγκτικές συνέδριες για τον ορίζοντα 2020 και εξετάσαμε τα ποσοστά σφάλματος τα οποία υπολογίστηκαν τόσο για το ε, FP7 όσο και για τον ορίζοντα 2020. Με χαρά μπορώ να σας ανακοινώσω ότι το 2018 λοιπόν το σύνολο των ε, λογαριασμών των κοινών επιχειρήσεων παρουσιάστηκε θετικά. Σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές των ετήσιων λογαριασμών, διαπιστώθηκε κανονικότητα και νομιμότητα σε όλους τους τομείς. Έτσι λοιπόν η γνωμοδότηση που εκδόθηκε ήταν θετική. Γνώμη χωρίς επιφύλαξη. Τώρα σε ό,τι αφορά το Fusion for Energy είχαμε δώσει έμφαση σε συγκεκριμένα στοιχεία και το ελεκτικό συνέδριο σημειώνει τα θετικά βήματα που έγιναν για να βελτιωθεί, η διαχείριση των λογαριασμών. Θέλουμε όμως να επιστήσουμε την προσοχή στην αύξηση του κόστους και στην ε, εφαρμογή υπό το ε, ETA. Όπως γνωρίζετε, το Νοέμβριο του 2016 εγκρίθηκαν νέα project ε, τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν την το επιχειρησιακό του σκέλος το 2025. Η ολοκλήρωση του σταδίου της κατασκευής αναμένεται για το 2035. Εδώ παρατηρήθηκε αύξηση του κόστου. Το Fusion for Energy έκανε υπολογισμούς 12 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα 6,6 δισεκατομμύρια που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο το 2010. Και εδώ υπάρχει αύξηση λοιπόν. Τέλος, τονίσαμε τους τομείς όπου επιδέχονται βελτίωσης. Του οποίους βασίστηκε και η γνωμοδότησή μας. Οι τομείς αυτοί αναφέρονται με λεπτομέρεια στην έκθεση και αφορούν επίπεδα εφαρμογής των έργων, τι συνεισφορές του ιδιωτικού τομέα, θέματα διοίκησης, ορισμένα θέματα οικονομικής διαχείρισης και άλλα οριζόντια θέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και προσβλέπω στα σχόλιά σας. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας αυτή. Θα δώσουμε το λόγο στον ε, Μπαρ Μπίμπεκ πρώτα απ' όλα να μας κάνει μια παρουσίαση για την κοινή επιχείρηση των ε, κυψελών καυσίμων. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ και τους, ε, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα της Επιτροπής ΚΟΝΤ που μας ε, δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε το θέμα αυτό. Τα επιτεύγματά μας ποια είναι. Και γιατί η Ευρώπη κάνει τόσο πολλά για τις κυψέλες καυσίμων και υδρογόνου. Το πρώτο απ' όλα έχουμε το θέμα της ανταγωνιστικότητας. Θέλουμε οι επιχειρήσεις μας να είναι στην αιχμή του δόρατος. Δεύτερο είναι θέμα ενεργειακής ασφάλειας. Εάν μπορούμε να παράγουμε περισσότερη ενέργεια εδώ τοπικά στην Ευρώπη, θα είμαστε πιο ανεξάρτητοι. Και το τρίτο βέβαια είναι προφανές, είναι θέματα βιωσιμότητας. Έχουμε πολύ αυστηρούς στόχους για το 2030 και θα μπορούσαμε και να αυξήσουμε τις φιλοδοξίες μας το 50-55%. Οπότε τα FCH οπωσδήποτε θα είναι μία από τις σημαντικές τεχνολογίες για την επίτευξη αυτών των στόχων. Γιατί η τεχνολογία αυτή δεν εκπέμπει ε, αέρια Μόνο υδρογόνο είναι το υποπροϊόν. Ε, μόνο, συγγνώμη, νερό είναι το υποπροϊόν. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε καθαρές μεταφορές, ε, καθαρή παραγωγή ενέργειας για θέρμανση και για ηλεκτρισμό, για να θερμάνουμε τα σπίτια και τα γραφεία. Θα πρέπει να μειώσουμε τη χρήση σπανίων πρώτων υλών και επίσης θα έχουμε δυνατότητα να αποθηκεύουμε ενέργεια για να μην έχουμε προβλήματα διακοιμάσεις στο δίκτυο. Έχουμε λοιπόν 150 επιχειρήσεις που εργάζονται προς την κατεύθυνση αυτή και 50% πρέπει να τονίσω είναι μικρομεσαίες. Το μεγαλύτερο τμήμα του προπολογισμού μας, περίπου το 30% δαπανάται για τις μικρομεσαίες. Επίσης έχουμε έρευνα για τη χρήση του υδρογόνου, έχουμε 80 ερευνητικά ιδρύματα στην Ευρώπη και φυσικά ανάμεσα σε όλα αυτά είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενέργεια λοιπόν μεταφορές και τα οριζόντια θέματα. Για παράδειγμα, τυποποίησης. Έχουμε 246 προγράμματα που στηρίζονται με 59 εκατομμύρια δημοσίου χρήματος και 935 εκατομμύρια ιδιωτικών επενδύσεων. Βλέπετε λοιπόν πολύ περισσότερα δίνει ο ιδιωτικό τομέα. Επίσης κάνουμε και μια μελέτη φέτος και ένα οδικό χάρτη για το υδρογόνο μέχρι το 2050 και καταλήξαμε στα εξή, ότι το τετρογόνο θα μπορούσε να συμβάλλει στο 24% τη τελική ανάγκη ενέργεια, μπορεί να παράγει 560 εκατομμύρια τόνων, μπορεί να παράγει τεράστιο ποσό εισοδημάτων και 5,4 εκατομμύρια θέσει εργασία μπορούν να προκύψουν στον τομέα αυτό. Αλλά δεν είμαστε μόνοι. Συνεργαζόμεθα με τον υπόλοιπο κόσμο. Αναφέρθηκε το θέμα αυτό και στο ανακοινοθέν του G20 του υδρογόνο θα παίξει μεγάλο ρόλο στην αποανθρακοποίηση της παραγωγής ενέργειάς μας. Ποια είναι τα κυριότερα στοιχεία. Ένα σημαντικό πρόγραμμα ήταν ε, η αξία του υδρογόνου σε ένα συγκρότημα νησιών ένα συγκρότημα νησιών όπου διαπιστώνουμε ότι μπορούμε έτσι να παραγάγουμε την ενέργεια για ε, να θερμάνουμε τα σπίτια, τα σχολεία και για τις μεταφορές με ενέργεια που παράγεται στα νησιά. Το 2016 συνεργαζόμεθα, αρχίσαμε να συνεργαζόμεθα με περιφέρειες. Τώρα με 92 για να μάθουν την τεχνολογία αυτή, πώς μπορεί να χρηματοδοτηθεί η παραγωγή της, να φτιάξουν τους οδικούς τους χάρτες για να φτάσουν εκεί και να εμπλακούν και οι τοπικές επιχειρήσεις. Οι περιφέρειες μας είπαν ότι για τα επόμενα πέντε χρόνια θέλουμε να επενδύσουμε 1,8 δις. Ποικίλει το επίπεδο φιλοδοξίας τους. Αλλά μερικές μεγάλες περιφέρειες ήταν πολύ πιο φιλόδοξες. Να μια συγκεκριμένη που είπε θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κοιλάδα του υδρογόνου. Είναι στη Βόρεια Ολλανδία θα έχουμε λοιπόν την πρώτη κοιλάδα υδρογόνου, σαν την κοιλάδα πυρητίου, το Silicon Valley της ε, Καλιφόρνια. Η κοιλάδα λοιπόν υδρογόνου θα είναι στην, ε, η πρώτη στη Βόρεια Ολλανδία. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν και άλλες. Επίσης, κάποιες περιφέρειες είπαν ότι θέλουν ε, να συνεργαστούν για να πάνε πιο γρήγορα. Έχουμε λοιπόν 40 περιφέρειες που έχουν λοιπόν αυτή την εταιρική σχέση για τις κοιλάδες υδρογόνου με επικεφαλής την Βόρεια Ολλανδία, την περιοχή Ροδανού Άλπαιων και την Αραγών. Θέλουμε λοιπόν να υπάρξει ανταλλαγή εμπειριών για να επιταχύνουμε την ε, εφαρμογή για την παραγωγή υδρογόνου. Έχουμε 32 προγράμματα, 140 εκατομμύρια από το 2011 βλέπετε στις κόκκινες κοιλίδες έχουμε επιτύχει μείωση του κόστους και αύξηση της ε, χωρητικότητας. Τώρα είμαστε σε κλίμακα μέγα βατ, ίσως να περάσουμε και σε γίγα βατ. Από πέρυσι διαπίστωσαν οι επιχειρήσεις ότι χάρη στην έρευνα έχει μειωθεί το κόστος και έχει αυξηθεί το δυναμικό. Μεγάλες επιχειρήσεις όπως ε, Χαλιβουργίες και η Shell αξιοποιούν αυτή την τεχνολογία για να δημιουργήσουν πράσινο υδρογόνο. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι το υδρογόνο που παράγεται είναι πράσινο. Γι' αυτό έχουμε αυτές τις εγγυήσεις προέλευσης. Βλέπετε εδώ με τα διάφορα χρώματα πώς φαίνονται όλα αυτά. Έχουμε μια συμφωνία με τον κλάδο και για τους ορισμούς. Είμαστε ηγέτες, είμαστε στην πρωτοπορία, είμαστε τρία χρόνια μπροστά χάρη στην έρευνά μας εδώ βλέπετε πώς προχωράμε. Είμαστε πολύ καλύτεροι από την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να διατηρήσουμε την πρωτοπόρο θέση μας και γι' αυτό και ο κλάδος προτείνει αυτή την επιχείρηση παραγωγής 40 γιγαβάτ που θα επιτευχθεί χάρη στις καινοτομίες μας για τις μεταφορές. Όλα τα μέσα μεταφορών προσπαθούμε να τα επηρεάσουμε για παράδειγμα, έχουμε τα λεωφορεία με κυψέλε καυσίμων. Από το 2010 ασχολούμεθα με 1,8 εκατομμύρια ευρώ, χάρη σε όλη την έρευνα. Μειώσαμε το κόστος στα 500 εκατομμύρια. Έχουμε 12 εγχειρήματα τέτοιου τύπου λεωφορείων και φέτος για πρώτη φορά λάβαμε και ένα βραβείο ένα από τα λεωφορεία μας, η βελγική επιχείρηση Φανχόλ, πήρε το βραβείο για το καλύτερο για το καλύτερο λεωφορείο του χρόνου. Ναι, ε, συνεργαζόμαστε και με το ΣΕΦ. Έχουμε μια μεγάλη πρωτοβουλία για τα λεωφορεία υδρογόνου που μείωσαν το κόστος. Είναι σαν ε, το κόστος ενός λεωφορείου με, υβριδικού με δίζελ. Από το 2016 έχουμε ξεκινήσει και τις υποδομές και εδώ ηγούμεθα. Επειδή ξεκινήσαμε πρώτοι, από το 2006, έχουμε τόση πείρα που βοηθάμε άλλα τμήματα του κόσμου, την Καλιφόρνια, την Κορέα, την Ιαπωνία, να φτιάξουν τα κέντρα επαναφόρτισης. Η Δανία ηγείται σε αυτή την προσπάθεια. και έτσι δημιουργούμε θέσεις εργασίας και εξαγωγές. Φιλοδοξία μας είναι το 2025 να έχουμε 800 τέτοιους σταθμούς ανεφοδιασμού. Πολλά πρέπει να γίνουν για τη θέρμανση και ψήξη να, έχετε, θέλουμε, μια μικρή κλίμακα σε κατάσταση που να μπορείτε να βάλετε στο σπίτι σας για να παράγετε θέρμανση και ψήξη. Έχει γίνει πολλή έρευνα. Τώρα αρχίζουν να αναλαμβάνουν ε, την προσπάθεια οι κυβερνήσεις μέσω επιδοτήσεων. Έτσι μπορούμε να αυξήσουμε την κλίμακα. Για την ασφάλεια. Εκπαιδεύουμε τους πυροσβέστες. Αν γίνουν ατυχήματα με το υδρογόνο θα πρέπει οι πυροσβέστες να ξέρουν πώς να τα αντιμετωπίσουν και εστιάζουμε και στην εκπαίδευση. Εργαζόμεθα με μικρά παιδιά και 15 ετών, αλλά και ανθρώπους που έχουν πάρει κάποια διπλώματα ε, επαγγελματικά για να ξέρουν πώς να αξιοποιήσουν αυτή την τεχνολογία. Έχουμε επίσης ε, ένα δίκτυο που μας επιτρέπει να βοηθάμε οποιουσδήποτε θέλουν να εργαστούν σε αυτό το τομέα. Έχουμε και δραστηριότητες ενημέρωσης του ευρύτερου κοινού Βλέπετε ότι πηγαίνουμε, τους δείχνουμε αυτά τα οχήματα, τους δείχνουμε τους σταθμούς ε, αναφόρτησης και στη Δυτική και στην Ανατολική Ευρώπη. Και η Ανατολική Ευρώπη πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζει αυτή την τεχνολογία. Αυτές οι δραστηριότητες βοηθούν ακριβώς να υπάρξει συνειδητοποίηση. Συνεργαζόμαστε επίσης με άλλα ευρωπαϊκά μέσα χρηματοδότησης, κάνουμε διάφορες μελέτες, για παράδειγμα το shift to rail, να περάσουμε στους σιδηροδρόμους. Κάναμε κάποιες μελέτες για να δούμε πώς μπορούμε να συγχρηματοδοτήσουμε πρωτοβουλίες. Και επίσης με τους καθαρούς ουρανούς, Clean Sky, θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την τεχνολογία και για την κίνηση αεροπλάνων. Και εδώ θέλουμε κάποια κοινά εγχειρήματα να υπάρξουν. Άλλη κοινή προσπάθεια, με το ΣΕΦ. Κυκλοφορούν 125 τέτοια λεωφορεία όπου οι υποδομές πληρώνονται από το ΣΕΦ και η κοινή επιχείρηση πληρώνει τα λεωφορεία. Ο συνδυασμός εθνικών πόρων, περιφερειακών πόρων, του ΣΕΦ και των εγχειρημάτων μας, όλα αυτά βοηθούν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, αποτελέσατε πραγματική πρόκληση για τους ε, διερμηνείς αλλά βλέπω τον ενθουσιασμό με τον οποίο μας παρουσιάσατε τις ε, κοινέ επιχειρήσεις. Δεν ήθελα να σας διακόψω, λυπάμαι που το έκανα. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Σώμα και να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Γιωχάνες Σβέμερ και είμαι διευθυντής της κοινή επιχείρησης Σύνδεξη για την Παραγωγή Ενέργειας. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα εδώ πέρα και σε ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να σας εξηγήσω την πρόοδο που έχουμε σημειώσει στα πλαίσια της δημιουργίας του Διεθνούς Θερμοπυρηνικού Πειραματικού Αντιδραστήρα Twitter και είμαι προφανώς στη διαθεσή σας του τέλους παρουσιαστής μου για να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις. Αναφερόμαστε εδώ πέρα στην έμφαση επί ειδικού θέματος που αναφέρεται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο μας έδωσε μια θετική γνώμη, χωρίς επιφύλαξη δηλαδή, σας ευχαριστούμε γι' αυτό, και αναφερθήκατε βέβαια στην πολυπλοκότητα του όλου έργου ITER, καθώς επίσης και στην πολύ μεγάλη κλίμακα του έργου αυτού. Πάντως χαιρόμαστε πάρα πολύ για την θετική γνώμη χωρίς επιφύλαξη, την οποία χορήγησε το Ελεκτικό Συνέδριο. Περιμένουμε το 2035 να ολοκληρώσουμε τη φάση κατασκευής βάσει του τρέχοντος χρονοδιαγράμματος και έχει δίκιο το ελεκτικό συνέδριο όταν λέει ότι στο παρελθόν είχαμε πει ότι η καταληκτική ημερομηνία ήταν το 2020. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι οι συνεισφορέ προ την φάση οικοδόμηση δεν περιλαμβάνουν τις έκτατες εισφορέ. Το Brexit σίγουρα θα μα επηρεάσει. Παρ' όλα αυτά είμαστε πεπισμένοι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα, συνεχίσει με τον ένα τον άλλο τρόπο να συμβάλλει στο έργο αυτό. Επομένω, η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασίλειου από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα θέσει ένα αμφιβόλο ή ένα κινδύνο το έργο αυτό. Λέμε επίση ότι πολλά θα εξαρτηθούν όσον αφορά τι εισφορέ από το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Κάνουμε λοιπόν έκκληση προ όλου να συνεχίσουν να συνεισφέρουν στο έργο αυτό, προκειμένου να καταφέρουμε να το ολοκληρώσουμε μέχρι το 2027. Λέγεται επίση στην έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου ότι υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι σε σχέση με την αύξηση του κόστου και πιθανέ καθυστερήσει. Καταλαβαίνετε ότι αυτό Όντω προκύπτει φυσιολογικά σε ένα τέτοιο έργο, ενό τέτοιου μεγέθους. Παρ' όλα αυτά καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο αυτό και να μειώσουμε τους κινδύνους και τι καθυστερήσει. Τώρα, τι ακριβώς προσπαθούμε να πετύχουμε. Θυμάμαι την πρώτη φορά που είχα να σα δω, η κυρία Γκρέσλε τώρα προείδρευε, και μιλούσαμε για διάφορα επιστημονικά δεδομένα και μου είχε πει η κυρία Γκρέσλε τότε, σας παρακαλώ πολύ πείτε μου πραγματικά που πηγαίνουν τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Προσπαθούμε να κτίσουμε ένα μηχάνημα, το TOCMAC, όπου βλέπετε ότι προσπαθούμε να περάσουμε τα στοιχεία του πλάσματος στον αντιδραστήρα αυτό και προχωρούμε σε μια διαδικασία καύσης του πλάσματος προκειμένου να δημιουργηθεί θέρμανση και κατ' επέκταση ενέργεια. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να προκληθεί η καύση αυτή την οποία θέλουμε να δημιουργήσουμε και είμαστε πεπισμένοι ότι ο ΙΤΕΡ θα επιτύχει το στόχο αυτό. Να σε υπενθυμίσω ότι είναι το πλάσμα. Ξέρετε ότι το σύμπαν αποτελείται από πλάσμα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ουσιαστικά από αυτό απαρτίζει το ίδιο ο ήλιος ή τα αστέρια και ουσιαστικά είναι η μεγαλύτερη πηγή ενέργειας στο σύμπαν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν και τους ανθρώπους να καταφέρουν να συλλέξουν και να αποθηκεύσουν και να αξιοποιήσουν αυτή την πηγή ενέργειας. Αυτή τη στιγμή κάνουμε περισσότερη ενέργεια παρά τόσο ανάπτυξη στο έργο αυτό. Προσπαθούμε ακόμα να καταλάβουμε πώς λειτουργεί η ενέργεια αυτή. Πάντως σαφώς ε, προωθούμε συγκεκριμένες ιδέες για το πώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη σημαντικότατη αυτή πηγή για την παραγωγή ενέργειας στο μέλλον. Προκειμένου να το κάνουμε όμως αυτό θα πρέπει να δημιουργήσουμε όπως βλέπετε μια τεράστια εγκατάσταση, στη Νότια Γαλλία βρίσκεται αυτή, να εικόνα πριν από ένα χρόνο και να πως έχει το εργοτάξιο αυτό τον προηγούμενο μήνα, τον ε, Νοέμβριο. Πρέπει βέβαια να βάλουμε και μία στέγη και ήδη σήμερα το πρωί υπάρχουν κάποια τμήματα του εργοταξίου αυτού που έχουν τροποποιηθεί. Βλέπετε λοιπόν ότι πετυχαίνουμε απτά αποτελέσματα. Πάνω από 2.000 άνθρωποι εργάζονται στο εργοτάξιο αυτό και πιστεύουμε ότι η επίτευξη πρόοδου και η ταχύτητα ολοκλήρωσης του εργοταξίου αυτού είναι πάρα πολύ σημαντική, εφόσον μιλάμε μάλιστα και για έναν πυρηνικό αντιδραστήριο. Εδώ, εδώ πέρα βλέπετε τα μαγνητικά πεδία που λειτουργούν, τα μαγνητικά ποινία μάλλον, που λειτουργούν στο πλαίσιο ενό τοροειδού μαγνητικού πεδίου. Βλέπετε τα μαγνητικά βία αυτά καθεαυτά, πώ έχουν εγκατασταθεί και πώ συνδέονται με τα υπόλοιπα τμήματα. Βλέπετε πάλι την εικόνα τον περασμένο Νοέμβριο και πώ έχει τώρα η κατάσταση τον προηγούμενο μήνα. Βλέπετε εδώ πέρα ότι έχουν ε, μπει σε συγκεκριμένα χαλίβδινα πλαίσια, συνδέονται με τα υπόλοιπα, σύστημα, ε, τα υπόλοιπα τμήματα του συστήματος αυτού και καταλαβαίνετε ότι η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε για τη σύνδεση αυτή χρησιμοποιείται και σε άλλες εφαρμογές στη συνέχεια. Έχουμε έπειτα τα, τους υπόλοιπους μαγνήτες που γυρίζουν γύρω-γύρω από το σύστημα αυτό. Μιλάμε για τους πολοειδείς μαγνήτες, τα πολοειδή μαγνητικά ποινία. Έτσι είχαν τα πράγματα το Φεβρουάριο του 2017, όπου είχαμε κάνει μόνο μία εγκατάσταση για τα μαγνητικά αυτά ποινία, πάντα στο, στη Νότια Γαλλία. Ξέρετε ότι 300 περίπου τόνους ζυγίζουν τα ποινία αυτά, δεν μπορούσαν εύκολα να μεταφερθούν και τώρα βλέπετε πώς έχουν τα πράγματα τον προηγούμενο μήνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και στην εγκατάσταση αυτή σημειώνουμε πρόοδο. Τώρα, όσον αφορά την ευρύτερη προσέγγιση, μια συγκεκριμένη συνεργασία που έχουμε με την Ιαπωνία, που καταδεικνύει πραγματικά ότι με τη συνεργασία αυτή μπορούμε να χτίσουμε το τόκο ΜΑΚΑ. Έχουμε εδώ πέρα ένα μηχάνημα το οποίο φέρει την ονομασία JT60SA, το οποίο αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας με την Ιαπωνία. Βλέπετε πώς το μηχάνημα αυτό ήταν πριν από ένα χρόνο και πώς είναι τώρα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν και σε σχέση με το σχέδιο αυτό τα αρχικά μας σχέδια. Και βλέπετε εδώ πέρα του όντω μέσω της διεθνού συνεργασίας μπορούμε να χτίσουμε, να οικοδομήσουμε τέτοια μηχανήματα, τέτοια τόκομάκα. Οι επενδύσεις αυτές που κάνουμε είναι πάρα πολύ σημαντικές γενικότερα για τον κλάδο της κοινοτομία και της βιομηχανίας στην Ευρώπη. Ξέρετε ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικές συνεισφορές και συνεισφορές σε είδος όσον αφορά τον ίτερ. Υπάρχει μια ισότιμη κατανομή των συνεισφορών αυτών ανά την Ευρώπη και βλέπετε ότι συνεχώς επενδύουμε προς το όφελος της ευρωπαϊκής καινοτομίας για όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Και βλέπετε ότι υπάρχει μια έντονη καθαρή προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλα τα χρήματα τα οποία επενδύονται πραγματικά επηρεάζουν πολύ θετικά εν γέννη την ευρωπαϊκή οικονομία και τις υποδομές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακριβώς επειδή οτιδήποτε επενδύουμε ουσιαστικά αντιστοιχεί έπειτα σε καινοτόμες τεχνολογίες. Συμβάλλουμε λοιπόν πάρα πολύ εν γέννη στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό τομέα. Εποφελούνται πολλές επιχειρήσεις. Το ίμιση των χρημάτων βέβαια πηγαίνει αυτή τη στιγμή στην κατασκευή, στη φάση κατασκευής του ΙΤΕΡ συμμετέχουν πολύ μεγάλες ε, επιχειρήσεις αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδίως όσον αφορά τις α, ε, τεχνολογικές εξελίξεις. Τα μαγνητικά ποινία, τα οποία είδατε πριν από λίγο, ουσιαστικά έχουν δημιουργηθεί από τέσσερις μικρότερες τεχνολογικές επιχειρήσεις. Είχαμε και ένα εργαστήριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον προηγούμενο Ιανουάριο, όπου θυμάστε τότε ότι είχαμε καλέσει πολλούς εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας ε, που είχαν εξηγήσει τότε στους παρευρισκόμενους ευρωβουλευτές ότι ε, μιλάμε πραγματικά όχι για μία απλή θέση απασχόλησης, αλλά ουσιαστικά για επενδύσεις βιομηχανικές οι οποίες καθιστούν την Ευρώπη πιο ανταγωνιστική στο παγκόσμιο προσκήνιο. Εν κατακλείδη χαιρετίζουμε την γνώμη χωρίς επιφύλαξη του ελεγκτικού συνεδρίου. Το 2018 ήταν ένα έτος πολύ σημαντικών εξελίσεων. Βλέπετε ότι όντως μπορούμε να επιδείξουμε πλέον απτά αποτελέσματα και έχουμε κάποιες τροποποίησεις στο αρχικό μας σχέδιο κάθε τρεις ή τέσσερις μήνες. Η συνεργασία είναι πάρα πολύ καλή, ιδιαίτερα θετική συμμετέχουν πολλά ευρετικά ιδρύματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από όλες τις γωνιές του κόσμου προκειμένου να καταφέρουμε πραγματικά να διατηρήσουμε το αρχικό μας χρονοδιάγραμμα. Μπορεί όντω να έχουμε σημειώσει μια κάποια καθυστέρηση, παρόλα αυτά έχουμε επισπεύσει τις δραστηριότητές μας και έχουμε αρχίσει να προχωρούμε λίγο πιο γρήγορα και ενδεχομένω να καταφέρουμε τελικά να ολοκληρώσουμε τις, εγκαταστάσεις, τις εγκαταστάσεις των μαγνητών, των μαγνητικών ποινίων που σας έδειξα πριν από λίγο. Αυτό εξαρτάται όμω και από τη συνεργασία που έχουμε με την Ιαπωνία. Θεωρώ πάντω ότι καταφέρνουμε αυτή τη στιγμή και διασυνοριακά και διεθνικά να εργαζόμαστε πολύ γρήγορα. Α μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μια διάσταση διατήρηση τη ειρήνη, καθότι προσπαθούμε μέσω τη επένδυση αυτή να αποφύγουμε μελλοντικέ συγκρούσει. Όσον αφορά τον προπολογισμό, θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τα ανώτατα όρια του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου, μέχρι το 2020 και συνεχίσουμε να σημειώνουμε πρόοδο και στις εσωτερικές μας διαδικασίες με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Σας υπενθυμίζω ότι πριν από δύο χρόνια εορτάσαμε την δεκαετή μας επέτειο, επομένως ξεκινήσαμε από το μηδέν όσον αφορά το έργο για τη σύνδεξη για την ενέργεια, σημειώσαμε πρόοδο και θεωρώ ότι έχουμε αρχίσει να οριμάζουμε. Ολοκληρώνω στο σημείο αυτό και αναμένω τις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Σφέμα. Με αυτά που είπατε μου θυμήσατε τα πρώτα χρόνια που κάναμε τελείω διαφορετικές ερωτήσεις. Γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που τώρα έχουμε γίνει ακόμα πιο περίεργοι. Θέλουμε να μαθαίνουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα και αυτό έχει μεγάλη διαφορά από τότε, από την αρχή. Γι' αυτό λοιπόν σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και γι' αυτό που μα είπατε τώρα. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον ε, συναδέλφο που θα μα μιλήσει για τον ε, καθαρό ουρανό. Και είμαι πολύ, πολύ περίεργη να δω τι έχει να μα πει για την συνεργασία μεταξύ σας διότι η αεροπορική βιομηχανία είναι μία από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης και ε, με ενδιαφέρει να μάθω τι γίνεται ιδιαίτερα σε θέματα χρηματοδότησης. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Άξελ Κάιν και μετά στη Μαρτίνα, αν δεν κάνω λάθος. presentation seems to be not up yet. Δεν νομίζω πως είναι έτοιμη ακόμα η παρουσίαση. Θα περιμένουμε λίγο. Ωραία, θα, θα ξεκινήσω. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε σε αυτήν την συνεδρίαση. Είμαι καινούριο σχετικά στη θέση, γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα αυτής εξ αρχής να πω πως εκτιμώ πάρα πολύ την επικοινωνία που υπάρχει, με το Κοινοβούλιο και είναι η πρώτη συνεδρίαση που συμμετέχω και συζητούμε θέματα απαλλαγής. Καθαρός ουρανός 2, λοιπόν, περί τίνος πρόκειται. Αν περάσουμε στη δεύτερη σελίδα της παρουσίασης, είναι πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση πάντως, το ξέρετε. Και η προηγούμενη παρουσίαση είναι πάρα πολύ καλή. Εντάξει, αν μπορείτε να τη διαβάσετε, έχετε εξαιρετική όραση. Λοιπόν, η κοινή επιχείρηση Clean Sky, όπως γνωρίζετε, αποτελείται από τέσσερα δισεκατομμύρια και ταυτόχρονα εξετάζει θέματα ανταγωνιστικότητας και κινητικότητας. Βλέπετε στα αριστερά τους κύριους στόχους μας σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, ε, δηλαδή θέλουμε μείωση 20-30% διοξιδίου του άνθρακα, 20-30% μονοξίδιο του αζότου από τα ε, αεροσκάφη σε σχέση με το 2014, καθώς και μείωση της συγχωρήπανσης εστιάζουμε σε νέα διαμόρφωση των αεροσκαφών, νέες ιδέες για την κατασκευή, νέες ε, τεχνολογίες πρόσης και γενικότερα νεοτερισμούς έτσι ώστε να καταφέρουμε να εστιάσουμε στους στόχους και να τους επιτύχουμε. Σε ό,τι αφορά τους συμμετέχοντες τώρα, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ε, διαφών συμμετεχόντων από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βιομηχανία. Έχουμε περίπου 1.500 διαφορετικούς ε, συμμετέχοντες, διαφορετικές συμμετοχές σε 28 κράτη-μέλη σε όλη την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή Έχουμε φτάσει σχεδόν τις 500 επιχορηγήσεις που έχουν εγκριθεί και ε, χορηγηθεί στους δικαιούχους. Συνεργαζόμαστε με διάφορες ε, περιοχές της Ευρώπης, έχουμε κέντρα ε, διαχείρισης, χρησιμοποιούμε την ευφύ εξειδίκευση και παρέχουμε τεχνική στήριξη, βοήθεια στην αξιολόγηση και ε, συνδρομή στη χρήση των διαθροτικών ε, ταμείων σε θέματα αεροπλοείας. Περίπου το 70% της χρηματοδότησης του προγράμματος προέρχεται από ε, δημόσιους διαγωνισμούς. Έχουμε μεγάλη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες συμμετέχουν πρώτη φορά σε τέτοια προγράμματα πλαίσιο ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό είναι ενδεικτικό της ευκολίας πρόσβασης που υπάρχει για τις επιχειρήσεις αυτές και επίσης ε, τα ποσοστά επιτυχίας είναι αρκετά υψηλά ε, και οι επιχειρήσεις αυτές δηλαδή όταν κάνουν αίτηση χρηματοδότηση έχουν πραγματικές επιθανότητες να την λάβουν, έχουν ρεαλιστικούς στόχους. Τώρα, στηρίζουμε τις ε, προσπάθειες να πλαισιωθεί ε, τεχνολογικά η βιομηχανία και ε, ο στόχος είναι η ανάπτυξη αυτής. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεισφέρουμε σε αυτό. Τώρα υπάρχει ένα εύρος επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη. Στηρίζουμε σε όλες τις χώρες, όλα τα κράτη-μέλη επιχειρήσεις από την Ελλάδα ως την ε, Ιρλανδία. Είναι λοιπόν μεγάλη η συμμετοχή σε όλη την Ένωση. Να σας πω τώρα δύο λόγια για την ε, τεχνολογική πρόοδο. Έχουμε έξι χαρακτηριστικά παραδείγματα διαφορετικών προγραμμάτων. Στο πάνω μέρος έχουμε θέματα ε, πρόσης, έχουμε ε, προσπαθήσει να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα των ε, αεροσκαφών μικρής και μεσαίας εμβέλεια. Βλέπουμε τα, τα ζητήματα έτοιμο, τα επίπεδα ετοιμότητας μάλλον. Και ο τελικός στόχος είναι από το 2 στο 5. Είναι δηλαδή ρεαλιστική η στόχη. Θα δούμε για παράδειγμα το 2018 πιάσαμε έναν μεγάλο στόχο ε, στην αξιολόγηση και αναθεώρηση του, του σχεδιασμού και το 2021 θα γίνει η πρώτη έλεγχη στο έδαφος. Άλλες επιτυχίες του τομέα αυτού Έχουμε το TRL3, καμιά φορά φτάνει μέχρι και το 5 και στα δεξιά βλέπουμε την ε, αξιολόγηση του αρχικού σχεδιασμού το 2018 και τις προβλέψεις για το 2020 με στόχο δοκιμές ε, σε συνθήκες πτήσης το 2022. Στο κάτω μέρος βλέπετε την ε, καμπίνα, εξεκέλευτη καμπίνα πιλότου Προσπαθήσαμε εδώ να βελτιοποιήσουμε τις συνθήκες στην καμπίνα και για θέματα κόστους αλλά και για λόγους ασφαλείας. Και εδώ βλέπουμε ότι έχουμε πιάσει, ε, ότι ε, βλέπουμε τα ορόσημα μάλλον. Μετά, στο κάτω μέρος της σελίδας υπάρχει η, ε, υπάρχει, υπάρχουν οι αυτοπροσαρμοζόμενες πτέρυγες του αεροσκάφους. Προχωράμε σε πιο ηλεκτρικά αεροσκάφη έχουμε αντικαταστήσει τα παλιά συστήματα με ηλεκτρικά. Βλέπουμε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος και σε αυτούς τους τομείς. Τώρα σε ό,τι αφορά τα νούμερα. Κατά την ε, διαδικασία εκπόνησης της απαλλαγής. Έχουμε δει ότι οι πιστώσεις υποχρεώσεων και οι πληρωμών ε, έχουν φτάσει σχεδόν στο 100%, 100% για τις αναλήψεις υποχρεώσεων και 98,2% για τις επιστώσεις πληρωμών. Στο, κάτω μέρος της σελίδας βλέπουμε ότι υπάρχουν 1.228 εκατομμύρια, 1,2 δις δηλαδή, χρηματοδότηση της Ένωσης για τα μέλη. Και στο κάτω μέρος βλέπουμε 2,19 δις ιδιωτικές εισφορές σε είδος. Στα δεξιά του πίνακα αυτού βλέπουμε το τι έχουμε επιτύχει μέχρι στιγμής, μέχρι το τέλος του 2018, δηλαδή 507 εκατομμύρια χρηματοδότης Ευρωπαϊκής Ένωσης και 1,2 δις ε, ιδιωτικών εισφορών σε είδων. Υπάρχει λοιπόν ε, εδώ σημαντική πρόοδος. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ε, συνολικές προοπτικές, αν δούμε τις ε, συνολικές προοπτικές χρηματοδότησης, θα παρατηρήσουμε ότι υπάρχει μία καμπύλη αρκετά τυπική. Ξεκινάμε από το 2014 με αργούς ρυθμούς. Υπάρχει μία απότομη αύξηση και τώρα βρισκόμαστε στο τελικό ε, στάδιο των συστημάτων επίδειξης. Έχουμε περίπου το 43%, δαπανίσει το 43% των ε, πόρων και τώρα περνάμε στο επόμενο στάδιο, στο 65% δηλαδή στο ορόσημο των 2 τρίτων της χρηματοδότησης και Καθώς προχωράμε στην τελική φάση επίδειξης, έχουμε τον στόχο να καταφέρουμε να επιδείξουμε τις νέες αυτές τεχνολογίες, όχι μόνο δηλαδή ανάπτυξη, αλλά και επίδειξη σε συνθήκες πτήσης. Βλέπουμε λοιπόν ότι και εδώ στο, το 2021 θα φτάσουμε στο ανώτατα, στο ανώτατο σημείο και σιγά σιγά θα παρατηρείται μία μικρή στεδική μείωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά συστήματα ελέγχου, το ηλεκτικό συνέδριο ασχολήθηκε με θέματα χρηστής ε, οικονομικής ε, διαχείρισης. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που ακολουθήσαμε στο ηλεκτικό συνέδριο για τους εσωτερικούς ελέγχους εξετάστηκαν και οι εσωτερικές κανότητε ε, σε θέματα πληρωμών. Το ποσοστό σφάλματος βρίσκεται κάτω από το 2%, στο 1,2%. Αυτό μάλιστα το ποσοστό υπήρχε και από την ε, αρχή, από το ξεκίνημα του προγράμματος αλλά φροντίσαμε να μην ε, εξετάσουμε μόνο τα θέματα τεχνικά, εκτέλεσης, όμως και να υπάρχει ένα σύστημα χρηστής οικονομικής διαχείρισης. Τέλος, βλέποντας λίγο τις μελλοντικέ προοπτικές. Βλέπουμε, όπως είπε και ο συνάδελφος, ότι έχει ξεκινήσει συνεργασία με το SCH. Χρησιμοποιούμε το υδρογόνο για το μέλλον ε, και βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μεγάλη φιλοδοξία για, την, για να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050 ε, και δεδομένου του ψηφίσματος ε, που ενέκρινε το Κοινοβούλιο πρόσφατα για την κατάσταση περιβαλλοντικής έκτακτης ανάγκης, βλέπουμε ότι τώρα έχουν γίνει πολύ σημαντικά πρώτα βήματα που σίγουρα όμως ε, δεν αρκούν για να επιτύχουμε το στόχο μας. Το επιθυμητό είναι μια πραγματική τεχνολογική επανάσταση, όπως καταφέραμε και με τον Καθαρό Ουρανό 2. Θέλουμε να περάσουμε λοιπόν στην επόμενη φάση αλλά χρειάζονται ακόμα βελτιώσεις έτσι ώστε να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο. Χρειάζεται ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και γι' αυτό οφείλουμε να συνεργαστούμε πολύ στενά με τον Axel και, τις, ε, και το ε, ε, CFS. Έτσι ώστε να βελτιωπήσουμε την χρήση των πόρων για το στόχο αυτό που μας έχει δοθεί. Όπως σας είπα, δεν πρόκειται για εξέλιξη, δεν είναι εξέλιξη το ζητούμενο, είναι η επανάσταση. Και οι πρώτες ενδείξεις από τις συζητήσεις που είχαμε με τους ε, ιδιωτικούς φορείς είναι ότι υπάρχει η δυνατότητα, εάν ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας, από την πλευρά τόσο των αεροσκαφών όσο και των βιώσιμων καυσίμων, σε συνδυασμό με τις επιχειρησιακές βελτιώσεις να επιτύχουμε τον ε, στόχο για κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Αυτό όμως θα γίνει μόνο εάν ενώσουμε τις δυνάμεις μας και προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν μπορούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο στον συγκητή και μετά στη Ματίνα. Ευχαριστώ. Ε, με συγχωρείτε αλλά είμαι από την Ήτρε όπου συζητάγαμε μισό λεπτό, Μα και εγώ θέλω να ρωτήσω το Γενικό Διευθυντή Έρευνα. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε που πήρα το λόγο. Α, ευχαριστώ, είστε κύριος που μου αφήνετε να πάρω πρώτο το λόγο. Οι κοινέ επιχειρήσει για μένα πραγματικά αποδίδουν την προστιθέμενη αξία και πραγματικά είναι πρωτοπόρες στα πλαίσια του Horizon 2020. Δεν είναι απλώς ε, θέμα σωστής αξιοποίησης των πόρων, αλλά συνδυασμού δεξιοτήτων και γνώσης και για να γίνουμε πρωτοπόροι παγκοσμίω. Οι κοινέ επιχειρήσεις συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη. Είμαι, είμαι πεπισμένη και στη δημιουργία θέσεων εργασία. Πρέπει λοιπόν έτσι να αξιοποιήσουμε και να ενώσουμε διάφορες ε, που φαινομενικά άσχετες προσπάθειες. Αυτός είναι ο καλύτερος στόχος και θαυμάσια φιλοδοξία που επιτυχάνεται μέσω των κοινών επιχειρήσεων. Χαίρομαι λοιπόν που όλε οι κοινέ επιχειρήσει εξάγουν διδάγματα από τη μέχρι τούδε λειτουργία του. Με συγχωρείτε τα λέω γρήγορα γιατί δεν θέλω να σα καθυστερήσω. Χαίρομαι λοιπόν που όλοι βελτιώνονται μέσω της εμπειρίας τους γιατί εργάζομαι για τα θέματα αυτά, για τα θέματα αυτά εδώ και χρόνια και ξέρω ότι κάθε χρόνο τα πηγαίνουμε όλο και καλύτερα. Και η συνεργασία με το Λεκτικό συνέδριο μας βοηθάει. Υπάρχει διαφάνεια στη χρήση των ε, πόρων, για παράδειγμα, για τα έξοδα αποστολών. Βεβαίως χρειάζονται βελτιώσεις. Άρα να κάνω μερικές ερωτήσεις. Πρώτη προς το ελεκτικό συνέδριο. Είπατε ότι υπάρχουν μεθοδολογικές αδυναμίες όσον αφορά τον υπολογισμό του ποσοστού σφαλμάτων. Συζητήσατε με τις κοινέ επιχειρήσεις για να λύσετε το θέμα αυτό. Να υπάρχει μια ενιαία μεθοδολογία για όλους. Αν όχι, θα το κάνετε. Και πότε. Είναι δυνατόν να υπάρχει μια ενιαία μεθοδολογία και μία ερώτηση προς όλες τις ε, παρούσες κοινές επιχειρήσεις. Σύνδεξη για την ενέργεια. Δημόσιες προμήθειες. Βλέπω ότι το συνέδριο λέει ότι ο κίνδυνος για τις ε, δημόσιες προμήθειες είναι με τρίο επίπεδου. Τι θα κάνετε για να βελτιωθεί η κατάσταση. Πώς θα ε, εφαρμόσετε τα διδάγματα του παρελθόντος. Τρίτον, για το FCH. Θα ήθελα να μάθω τι έγινε με το 7ο επίπεδο εφαρμογής. Από την πείρα σας θεωρείτε ότι θα επαναληφθεί η κατάσταση ή στο νέο πρόγραμμα θα τα πάμε καλύτερα για να βελτιωθεί ε, το ποσοστό απορρόφησης και για τους καθαρούς ουρανούς και καλωσορίζω στην διαδικασία την τόσο συναρπαστική απαλλαγή σε αυτή την τόσο συναρπαστική επιτροπή μας τον νέο διευθυντή τον συγχαίρω για το επίπεδο εφαρμογής που είναι περίπου 100% για το FP7 το 2018 κάνατε ανακτήσεις 0,85 εκατομμυρίων ευρώ λόγω, λόγω προβλημάτων με την προχρηματοδότηση και με τους ελέγχους. Τι θα γίνει με αυτό το ποσό και τι μπορούμε να κάνουμε για να προλαμβάνονται τέτοιες καταστάσεις στο μέλλον. Αυτά και ζητώ συγγνώμη τον εισηγητή. Ο Μάρκος Πίπερ θα είναι μετά τον εισηγητή. Α, όχι, τελικά θα μιλήσει γιατί χρειάζεται να μιλήσει πρώτα ο Μάρκο Πίπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον εισηγητή. Ο κύριος εισηγητής, μα έχω κάθε κατανόηση για όλους. Σε ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Πίπα. Η, η προηγούμενη ήταν πιο έξυπνη από μένα και εκείνη πρέπει να πάει στην ε, ίδια ψηφοφορία με μένα, αλλά μίλησε πριν από μένα. Εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Τρία συντόμω. Πρώτον, με εντυπωσιάζει το πόσο καλά τα πάνε οι κοινέ επιχειρήσεις. Το ερώτημά μου είναι πώς θα πάει στις περιφέρειες αυτή η προστιθεμένη αξία, ούτω ώστε και οι πολίτες μας να ενημερωθούν καλύτερα πόσο θετικά πράγματα κάνουμε. Ότι είναι πραγματικά γνήσια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Και θεωρώ ότι ότι θα πρέπει να ενημερώσουμε την κοινή γνώμη, να την ευαισθητοποιήσουμε για αυτά μας τα επιτεύγματα. Δεύτερον, μικρομεσαίες. Είπατε ότι θέλετε να συμμετάσχουν περισσότερο. Πώς ακριβώς ε, συμμετέχουν, πού τις βρίσκεται. Γίνεται μία προκήρυξη που μπορεί μια μικρομεσαία επιχείρηση στην Αυστρία ή τη Γαλλία να μην την πάρει Γιατί δεν τα παίρνουν είδηση αυτά τα μεγάλα πράγματα. Πώς προκύπτουν, πού τις βρίσκεται αυτές οι μικρομεσαίες για να συμμετάσχουν στα προγράμματά σα για όλες τις ε, κοινέ επιχειρήσεις αυτά, για αυτή η ερώτηση. Και για τους καθαρούς ουρανούς. Με, με εντυπωσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας. Αλλά το ερώτημά μου είναι πόσο κοντά είμαστε στο τέλος. Θα καταφέρουμε να πετάνε αεροπλάνα με αυτές τις τεχνολογίες. ή θα υπάρχουν προβλήματα για να λειτουργήσει. Και κάτι ακόμη. Θέλω να εκφράσω την απογοήτευσή μου για το υδρογόνο. Κοιτάξτε, υπάρχουν ε, αεροσκάφη που πετάνε ήδη με υδρογόνο. Και εσείς λέτε ότι είναι μεγάλη πρόκληση του μέλλοντος. Εγώ θα νόμιζα ότι η τεχνολογία έχει ήδη προχωρήσει. Από ό,τι κατάλαβα από την παρουσία. ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος. Λοιπόν, ε, να απαντήσουν οι κοινές επιχειρήσεις του ώστε ο συγητής να μπορεί να κάνει ε, με την ησυχία του τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ, Γιωχάνες Φένε ανάπτυξη της ενέργειας από τη σύνδεξη. Να απαντήσω στην ερώτηση που έγινε κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πώς μπορούμε να τις εμπλέξουμε περισσότερο ώστε να αποφεληθούν και αυτές. Οι δημόσιες προμήθειες έχουν ουσιαστικά τρεις αν θέλετε κινδύνους. Πρέπει καταρχάς να βρούμε αναδόχους και πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Πώς μπορούμε να βρούμε πολλούς συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς και πώς μπορούν έπειτα οι επιλεχθέντες πραγματικά να ανταποκριθούν στο σχέδιο το οποίο πρέπει να επιτελέσουν. Συνεργαζόμαστε με το Aeroforum στα πλαίσια Twitter, με μεγάλα ερευνητικά ιδρύματα όπως ο Ευρωπαϊκός Διαστημικός Οργανισμός ή το CERN και προσπαθούμε ουσιαστικά κάθε δύο χρόνια να δημιουργήσουμε μεγάλα φόρουμ όπως το Big Science, το επόμενο θα γίνει για παράδειγμα στη Γρανάδα της Ισπανίας, συμμετέχει ο Ίτερ προφανώς και μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να φέρουμε από κοινού μεγάλες βιομηχανίες αλλά και ερευνητικά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με επιχειρήσεις και να τις πείσουμε τελικά ότι όντως αξίζει να συνεργαστούν με εμά για το project αυτό, για το έργο αυτό, μπορώ ότι παραδέχομαι ότι όλη η διαδικασία δημοσίων προμηθειών και σύναψη συμβάσεων είναι αρκετά πολύπλοκη και μπορεί τελικά να αποθαρρύνει κάποιες επιχειρήσεις. Έπειτα υπάρχει και το ζήτημα της ταχύτητας. Εμείς ξεκινήσαμε από μια διαδικασία που βασόταν σε κανόνε, μια διαδικασία που βασίζεται σε συγκεκριμένε πλέον διαδικασίε. Χρησιμοποιούμε τι νέε τεχνολογίε προκειμένου να καταφέρουμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Χρησιμοποιείται η ψηφιοποίηση επίση, προκειμένου μέσω τη ιστοσελίδα μα να μπορούμε να ερχόμαστε σε επαφή με επιχειρήσει και να βρίσκουμε τι απαραίτητε λύσει. Όσον αφορά έπειτα το κίνδυνο, όταν ήμασταν μικροί, αναζητούσαμε έναν μεγάλο ανάδοχο που θα μπορούσε να επιτελέσει όλα για μα. Τότε αισθανόμασταν αδύναμοι. Τώρα έχουν αντιστραφεί τα δεδομένα. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να συνεργαστούμε και με πιο, πιο μικρέ εξειδικευμένε επιχειρήσει για συγκεκριμένε συνιστώσει, με συγχωρείτε, για συγκεκριμένα εξαρτήματα θα έλεγα ότι ήταν πολύ πιο δαπανηρή η διαδικασία και πιο πολύπλοκη στην αρχή, αλλά καταλήγουμε τελικά αυτή τη στιγμή μια διαδικασία πολύ πιο γρήγορη, πολύ πιο αποτελεσματική. Και να περάσω κατά αυτόν τον τρόπο και στο άλλο ερώτημα, πώς βρίσκουμε και πώς προσελκύουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο περιθώριο των συνεδριάσεων αυτών συνεργαζόμαστε με τους λεγόμενους ILO officers. Υπάρχει ένα σε κάθε κράτος μέλος και κάθε κράτο μέλο αποφασίσει τελικά ποιο θα είναι το άτομο αυτό, πού θα βρίσκεται, πώ θα πληρώνεται. Έχουμε πάντω εμεί ένα δίκτυο με του ανθρώπου αυτού, γνωρίζουν ποιε είναι οι επικείμενε δημόσιε συμβάσει και ουσιαστικά αποτελούν ένα σύνδεσμο για αυτά τα κράτη-μέλη σε σχέση με τις βιομηχανικές αυτές σημαντικές εξελίξεις. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε μέσω των ILO officers να εμπλέξουμε περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλα τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ίσως ε, ο κύριος Κράνη και ο συνάδελφος ε, θα μπορούσαν να απαντήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω στην πρώτη ερώτηση για τον προϋπολογισμό. Έχουμε λοιπόν 1.500 ε, συμμετοχές και μετά την, τον έλεγχο τα ποσά αυτά θα μεταφερθούν στο επόμενο έτος. Αυτή είναι μια συνηθισμένη διαδικασία. Έχει κλείσει ήδη το θέμα, έχει ολοκληρωθεί, οπότε δεν υφίσταται πια. Η δεύτερη ερώτηση που έχει να κάνει με τις ε, δημόσιες σχέσεις για να ενημερωθεί ο κόσμος για αυτό που κάνουμε. Εμείς ε, φυσικά χρησιμοποιούμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να φτάσουμε στο ευρύ κοινό και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους. Πηγαίνουμε στα πανεπιστήμια τακτικά, έτσι ώστε να αυξηθεί το ενδιαφέρον των φοιτητών για αυτό που κάνουμε και ίσως ε, να τους ενδιαφέρει και έτσι ώστε να ακολουθήσουν κλάδους σπουδών στον τομέα αυτών. Επίσης, συμμετέχουμε σε συνέδρια σε όλη την Ευρώπη, έτσι ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες ε, για το τι κάνουμε. Τώρα, υπάρχει αρκετά μεγάλη συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η επιλογή τους γίνεται με κανονική διαδικασία αξιολόγηση από εμπειρογνώμονε. Τώρα, εμεί συμμετέχουμε σε τοπικέ εκδηλώσει που διοργανώνουν τα κράτη-μέλη, όπου καλούν εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πιθανότατα θα θέλουν να συνεργαστούν, τους εξηγούμε τα ωφέλη, τις τεχνικές λεπτομέρειε έτσι ώστε να τους κερδίσουμε. Αυτό κάνουμε τα τελευταία χρόνια και επίσης με τον τρόπο αυτό ε, αποκτούμε πρόσβαση και σε επιχειρήσεις που συνήθως δεν έχουν σχέση με την αεροπλοεία. Τώρα ε, η πρόσβαση στην αγορά αυτό εξαρτάται και από ε, τις δυνατότητες της τεχνολογικές. Τώρα βρισκόμαστε σε επίπεδο 6 σε συνθήκες πτήσης και μετά η εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής στο προϊόν έτσι ώστε να φαίνεται, ε, συμβαίνει 6 8 χρόνια αργότερα. Είναι τόσο το χρονικό διάστημα που χρειάζεται από τη στιγμή που μια τεχνολογία μέχρι τη στιγμή που θα την εφαρμόσει ένα προϊόν. Τώρα τα αεροσκάφη με υδρογόνο. Δεν υπάρχουν τέτοια αεροσκάφη που καίνουν υδρογόνο αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κάποια δοκιμαστικά αεροσκάφη, όμως ε, δεν ε, χρησιμοποιούνται σε εμπορικές πτήσεις. Αυτό οφείλεται εν μέρη στο γεγονός ότι το υδρογόνο είναι δύσκολο καύσιμο στο χειρισμό. Ιδιαίτερα για θέματα ασφάλειας. Για να πιάσει τα επίπεδα ασφάλειας που χρειάζονται ε, στην αεροπλοεία. Είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα και αυτό φαίνεται και από την ε, τωρινή κατάσταση με τις κυψέλες ε, υδρογόνου και καυσίμων. Εμείς συνεργαζόμαστε και με την ε, Brown έτσι ώστε να προχωρήσουμε την τεχνολογία αυτή και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ασφαλείας. Εστιάζουμε λοιπόν σε αυτό καθώς και στις ε, απαιτήσει για την αεροπλοεία. Για να σας δώσω μια εικόνα, ο όγκος του υδρογόνου είναι τρεις φορές μεγαλύτερος από εκείνον της κυροζήνης και αυτός ο όγκος είναι πολύ μεγάλος, πρέπει να ψυχθεί στους ε, μείον 250 βαθμούς για να γίνει υγρό, το οποίο παρουσιάζει πολλές προκλήσεις. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή κατάλληλη τεχνολογία έτσι ώστε να γίνει αυτό με ασφάλεια. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο Συνάδελφοι για την FCH. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του FP7, είμαστε στο 90% φέτος και μάλιστα φέτος ολοκληρώθηκαν πάρα πολλά έργα, τα οποία θα δείτε στην απαλλαγή για το, 2000, για το επόμενο έτος, το 2019. Υπάρχουν φυσικά κάποιες εκκρεμότητες, ε, από τις οποίες βέβαια αντλήσαμε διδάγματα. Ε, και πολλές φορές χρησιμοποίησαμε αυτά που μάθαμε στο παρελθόν και τα εφαρμόσαμε στον ορίζοντα 2020. Το ουσιαστικό και το βασικό για μας είναι να υπάρχει σωστός συντονισμός. Φυσικά, παρακολουθούμε και ελέγχουμε στενά την πρόοδο και επίσης ε, λειτουργούμε συμβουλευτικά και καθοδηγητικά τα προγράμματα του ορίζοντα 2020 τα πάνε πάρα πολύ καλά σε επίπεδα ε, εκτέλεση, οπότε δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα εδώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι περιφέρειε, ε, ιδιαίτερα τι εξόχω απόκεντε, ε, υπάρχουν ορισμένα έργα, για παράδειγμα τα λεωφορεία, τα ελαφρά λεωφορεία, τα οποία μπορούν να γίνουν αρκετά ορατά από τους πολίτες. Δηλαδή, όποιος χρησιμοποιεί ένα τέτοιο λεωφορείο, παθόρυβο, που δεν ρηπαίνει μπορεί να το διαπιστώσει από την πρώτη στιγμή. Υπάρχουν λοιπόν σε ορισμένες περιπτώσεις πάρα πολύ ε, ξεκάθαρα ωφέλη και μεγάλη ορατότητα. Αυτό που προσπαθούμε τώρα να κάνουμε είναι να συμμετέχουν όλοι οι πολίτες σε ένα έργο. Αυτό κάναμε στην Ολλανδία, αυτό κάνουμε και στις ε, Ορκάδες. Προσπαθούμε λοιπόν να αυξήσουμε την ορατότητα ενό ε, project, αυξάνοντα και τη συμμετοχή όλων των ε, πολιτών εκεί. Τα περισσότερα έργα επίσης ε, πρέπει να γίνουν τοπικά, πρέπει να ηγηθούν οι τοπικές κοινότητες στην διαχείρισή τους. Εμείς έχουμε διαφορετικό ρόλο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υπάρχουν αρκετές που συνεργάζονται μαζί μας και πώς τις βρίσκουμε αυτές. Νομίζω πως ε, αυτό γίνεται μέσω διαφόρων ενώσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω εθνικών σημείων επαφής. Εμείς πηγαίνουμε, όπως ε, σας είπα, σε πάρα πολλά συνέδρια, γι' αυτό ε, δεν υπάρχει ανησυχία για το ότι δεν μπορούν να μας βρουν αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, είμαστε πάρα πολύ ενεργοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Έχουμε λοιπόν ορατότητα τώρα σε ό,τι αφορά τα αεροσκάφη και το υδρογόνο. Εμείς εδώ και πολλά χρόνια μελετάμε τη χρήση υδρογόνου στην ε, αεροπλοεία σε διάφορα συστήματα, για παράδειγμα στην ε, θέρμα στην κουζίνα του αεροσκάφους, αλλά όχι ακόμα σε θέματα πρόσης. Το 2016 ξεκίνησαν κάποια, δοκιμασ... κάποια δοκιμαστική ε, κάποια δοκιμαστικά έργα, όμως ε, ακόμα δεν έχουμε περάσει σε εφαρμογή μεγάλη κλίμακα. Όπω σα είπε ο Άξελ, υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι και χρειάζεται ακόμα πάρα πολύ έρευνα, ε, ιδιαίτερα σε θέματα αποθήκευσης κρυογονική, του υδρογόνου, κάτι το οποίο δεν χρησιμοποιείται στις χερσαίες μεταφορές, οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα λοιπόν, επιτέλους να πάρει το λόγο και ο εισηγητής που θα έπρεπε να έχει μιλήσει πολύ νωρίτερα, αλλά σα ευχαριστώ πολύ για την κατανόησή σας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Επειδή με ενδιαφέρει η αγαστή συνεργασία με τους συναδέλφους, δεν είχα πρόβλημα να περιμένω λίγο. Γιατί καταλαβαίνω ότι οι συναδελφοί μου έχουν υποχρεώσει. Και ούτω ή άλλω οι απαντήσεις που δόθηκαν στι ερωτήσει που έκαναν οι συνάδελφοι καλύπτουν και δικέ μου ερωτήσει. Πρώτον, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι και κύριοι εκπρόσωποι των κοινών επιχειρήσεων, ευχαριστώ και την Πρόεδρο για τον πολύ αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ όλους και από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τις παρουσιάσεις σας και για τις επαφές που είχαμε πριν από τη συνεδρίαση που με επέτρεψαν να κατανοήσω τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο στην εργασία του. Είναι δυσχερή εργασία αλλά ιδιαίτερα σημαντική. Χάρη στην εργασία όλων αυτών κατάφερα να εκπονήσω κι εγώ τη γνωμοδότηση και τις ερωτήσεις μου. Υπάρχουν οκτώ κοινέ ευρωπαϊκέ επιχειρήσει στον χώρο τη έρευνα. Και πρέπει να χορηγήσουμε απαλλαγή και στι 8 για το 2018. Στο παρελθόν είχαμε χορηγήσει πάντα ε, απαλλαγή και χωρίς καθυστερήσεις. Την πρώτη φορά, που, η τελευταία μάλλον φορά που υπήρξαν προβλήματα ήταν το 2013 και το 2014, δηλαδή εδώ και αρκετά χρόνια. Το 2018 λοιπόν είχαμε τις γνωμοδοτήσεις ε, μέσω μιας ενιαίας έκθεσης ε, του ελεκτικού συνεδρίου και για τις οκτώ κοινέ επιχειρήσεις. Αυτό δεν αλλάζει την ουσία της διαδικασίας. Οι κοινέ επιχειρήσεις ε, πρέπει να λάβουν απαλλαγή όπως και οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί της Ένωσης. Όμως υπάρχει μια διαφορά. Αυτή το βασικό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι οι εκθέσεις του ελεκτικού συνεδρίου αναλαμβάνουν και όλες τις ε, συστάσεις ε, περιλαμβάνουν και όλες τις συστάσεις που δεν έχουν επιληθεί από προηγούμενες ε, απαλλαγές και δίνουμε απαλλαγή σε κάθε μία κοινή επιχείρηση, όχι γενικά, με βάση ακριβώς τη γνωμοδότηση του Ελεκτικού Συνεδρίου και διάφορα έγγραφα που αφορούν την οικονομική διαχείριση κάθε κοινή επιχείρηση, κάθε οικονομικό έτος. Έχουμε λοιπόν και την τελική έκθεση για τη χρήση του προπολογισμού και έχουμε και τις εκθέσεις δραστηριότητας των κοινών επιχειρήσεων αυτών. Οπότε, Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα τα οποία εντοπίζει το ελεκτικό συνέδριο. Η ετήσια έκθεσή του για τις κοινέ επιχειρήσεις δημοσιεύτηκε στι 14 Ιουλίου, όπου τονίζει το ελεκτικό συνέδριο ότι είναι αξιόπιστη οι λογαριασμοί των κοινών επιχειρήσεων και το ποσοστό σφαλμάτων για καμία κοινή επιχείρηση δεν υπερβαίνει το κατόφλιο του 2%. Ναι, μεν ε, καθυστερεί η εφαρμογή του, 2000, ε, του 2020 και αυτό δεν μας ικανοποιεί. Και ιδιαίτερα για το ITER και το FCS υπάρχουν καθυστερήσεις. Οι τρεις κοινέ επιχειρήσεις που προσκλήθηκαν εδώ σήμερα, η πρώτη είναι το FCH, εδώ ο έλεγχος του ελεκτικού συνεδρίου είναι θετικός. Δεν υπάρχουν μεγάλων ε, διαστάσεων προβλήματα. Είναι μια επιτυχημένη λοιπόν σύμπραξη ιδιωτικού δημόσιου τομέα. Η ερώτησή μου είναι κατά αυτήν την προγραμματική περίοδο. Πώς συνεργάζεστε με τον ορίζοντα 2020. Πόσοι χρειάζεται να εργαστούν για την απαλλαγή, πόσο κοστίζει. Η γραφειοκρατία είναι ανάλογη ή δυσανάλογη. Θεωρείτε ότι είναι καλό παράδειγμα σύμπραξης ε, δημοσιοδιωτικού τομέα λοιπόν αυτή για το FCH. Ένας από τους διευθυντές είπε κάτι που θέλω να σχολιάσω. Ότι συλλέγεται τεράστια επιστημονική γνώση. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτό βεβαίως και εμείς εκτιμούμε ότι είναι ιδιαίτερα πολύτιμο, αλλά ο ρόλος μας εδώ ως επιτρομή, Επιτροπή είναι να καταλάβουμε εάν ε, δαπανάτε σωστά ο προπολογισμό σας. Πρέπει να ελέγξουμε κάθε ευρώ του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε ότι δημιουργούνται τεχνολογίες, ε, Όμως, το πιο σημαντικό για μας είναι η χρηστή οικονομική διαχείριση. Τώρα, το f 4 e η σύνδεξη για την ενέργεια, είναι το πιο περίπλοκο, είναι πραγματικά τεραστίων διαστάσεων εγχείρημα. Υπάρχουν κάποια σημεία που θα πρέπει να τα δούμε. Το σημείο 3 για παράδειγμα. Η έκθεση λέει ότι αυξάνονται οι εισρωές. Το κόστος του δηλαδή. Πώς σχετίζεται αυτό με αυτό που αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και στο 4 λέμε ότι υπάρχουν πρόοδοι για το πλάσμα και λέτε ότι θα ολοκληρωθεί το 2025 η φάση οικοδόμησης. Στην παράγραφο 1 λέτε ότι υπάρχουν κίνδυνοι που συνδέονται με τον Brexit. Επίσης, ε, το Συμβούλιο Ευρατόμ παίζει σημαντικό ρόλο για το ίτερ συνολικά από το 2020 και μετά. Κατόπιν. Παράγραφος 10. Εδώ λυπούμεθα που δεν τηρήθηκε ο προπολογισμός. Υπήρξε υπέρβαση του προπολογισμού το 17-18 σε σχέση με τον αρχικό προπολογισμό. Αυτό είναι λυπηρό. Παράγραφος 20. Εσωτερικές στρατηγικές επικοινωνίες δεν επετέχθησαν. Θα παρακαλούσα τον Διευθυντή να αναφερθεί σε όλα αυτά τα σημεία. Τέλος. Καθαρή ουρανή 2. Όπως και για το FCH είναι θετικό το αποτέλεσμα του συνεδρίου, δηλαδή η εκτίμησή του. Ερώτηση ωστόσο, πώς θα συνεργαστείτε σε αυτή τη φάση προγραμματισμού με τον ορίζοντα 2020. Κατά λίγο λοιπόν και σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ λέει και η Πρόεδρος. Να δώσω το λόγο στη σκιώδη η κυρία Γκραπίνη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ελπίζω ότι θα είμαι πιο σύντομη από τον εισηγητή, ο οποίος έκανε μια πολύ ε, λεπτομερή παρουσίαση. Θα ήθελα καταρχάς να χαιρετήσω και εγώ τα θετικά αποτελέσματα από τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα θετικά πολλά αποτελέσματα που έχουμε για τις κοινέ επιχειρήσεις είναι σαφή τα αποτελέσματα όσον αφορά την νομιμότητα και την κανονικότητα των ετησίων λογαριασμών. Αυτό μας ενδιαφέρει εδώ πέρα, το είπε και ο εισηγητής, μας ενδιαφέρει να επενδύεται αποδοτικά το παραμικρό ευρώ του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Θα θέλαμε λοιπόν να δούμε την τάση αυτή τη θετική να συνεχίσετε και στο μέλλον. Παρόλα αυτά, το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο σε κάποιου τομεί έχει εντοπίσει ένα περιθώριο βελτίωση για να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. Περιμένουμε λοιπόν ότι οι κοινέ επιχειρήσει θα λάβουν υπόψη του τις συστάσεις αυτές και μέσω του εγχειρή, της απαλλαγής θέλουμε και εμείς να παρακολουθήσουμε πώς εφαρμόζονται αυτές οι συστάσεις. Σας παρακαλώ μιλήστε λίγο πιο αργά. Έχουμε ακόμα δύο λεπτά. Σαφώς. Καταρχάς, να θέσω κι εγώ κάποια ερωτήματα. Στην ετήσια έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο μας λέει ότι στα τέλη του 2018, στα μέσα δηλαδή της προγραμματικής περίοδου, οι 7 κοινέ επιχειρήσεις που εφαρμόσουν τις δραστηριότητες του ορίζοντα 2020 εφάρμοσαν ένα πολύ μικρό ποσοστό μόνο, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι θα πρέπει να ήταν 60% στα τέλη του 2018 το ποσοστό εκτέλεσης. Πώς εξηγεί εδώ πέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αντιστοιχία ανάμεσα στο ποσοστό εφαρμογής και το ποσοστό εκτέλεσης. Να αναφερθώ τώρα σε δύο κοινέ επιχειρήσεις και στις παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στην αφορά τις εισίδωσης φορές. Εδώ έχουμε ένα ποσοστό εκτέλεσης 25%. Πώς εξηγείται αυτό. Τρίτη ερώτηση. Για το JU, την κοινή επιχείρηση ενέργεια από τη σύνδεξη, για το 2017 και τη σχετική απαλλαγή είναι θετικά τα αποτελέσματα σίγουρα, αλλά έχετε κάποιο σχέδιο δράσης για τον αντίκτυπο που θα έχει το Brexit όσον αφορά τον θερμοπυρηνικό πειραματικό αντιδραστήρα. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Ριβαζή και μετά στον κύριο Κούς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ομολογώ ότι εγώ είμαι πολύ πιο σκεπτική σε σχέση με τις παρουσιάσεις αυτές. Αν πάρουμε το 2018 μας λέτε όλα πάνε πολύ καλά, καταπληκτικά. Όταν όμως βλέπω το σχέδιο σύνδεξης Twitter, νομίζω ότι εδώ πέρα θα πρέπει να διαρευνήσουμε λίγο περισσότερο την κατάσταση. Γιατί αν δούμε την περίοδο 2007-2027, ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό ζητήθηκε τουλάχιστον. Με όλες αυτές τις αβεβαιότητε και αναφερθήκατε και στο Brexit και ξέρουμε είτε πρόκειται για το Brexit με συμφωνία ή όχι, το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει σε κάθε περίπτωση από το Ευρατόμ. Θα έχουν όμω το καθεστώ τη Ελβετία. Αν δεν έχουμε συμφωνία αποχώρηση, δεν θα έχουν το καθεστώ Ελβετία οι Βρετανοί. Και Α μην ξεχνάμε ότι η Αγγλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, συμμετείχε στην πρόσκληση υποβολή προσφορών. Τι θα γίνει με αυτό στο μέλλον, δεν θα έχουμε εδώ πέρα καθυστερήσει. Δεν ξέρω αν το συνειδητοποιείτε σε σχέση με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, όπου θα πρέπει ουσιαστικά οι επενδύσει να είναι αποδοτικέ και αποτελεσματικέ. Το σχέδιο αυτό που θα έπρεπε τουλάχιστον στην πρώτη φάση για το πλάσμα να ολοκληρωθεί μέχρι το 2020, μα λέτε τώρα θα πρέπει να πάτε μέχρι το 2035. Και το σχέδιο αυτό έχει να κάνει μόνο με το πλάσμα αυτή τη στιγμή και στην Γαλλία ξέρετε ότι λέμε ότι πρόκειται για τον πιο ακριβό οργασμό ουσιαστικά, γιατί θα έπρεπε ουσιαστικά το πλάσμα αυτό να, να αποδώσει πάρα πολύ ενεργητικά. Θα πρέπει να φτιάξουμε όχι μόνο έναν, ένα δεύτερο αντιδραστήρα και θα απαιτηθούν και άλλε τεχνολογικέ εξελίξει για να καταφέρουμε τελικά να αξιοποιήσουμε την επένδυση αυτή. Το θέλουν αυτό οι πολίτε όμω. Αυτή τη στιγμή κάνουμε επενδύσει πολύ δαπανηρές, μας δείξετε και μια εικόνα του ήλιου και της ηλιακής ενέργειας. Το πρόβλημα όμως είναι ότι αν πραγματικά υπάρξει κάποιο πρόβλημα, δεν θα, δεν θα καταφέρουμε να τα βγάλουμε πέρα, δεν θα καταφέρει να αντέξει το όλο αυτό εγχείρημα σημαντικέ αλλαγέ ή απειλέ που μπορεί να έχουμε στο μέλλον. Γι' αυτό το λόγο και ω έχω, Γαλλίδα έχω πάρα, πάρα πολλού ενδιασμού όσον αφορά το ίτερ. Υπάρχουν πάρα πολλοί θειασότε του προγράμματο αυτού που λένε πω θα πάμε καταπληκτικά, θα εκμεταλλευτούμε την ηλιακή ενέργεια. Υπάρχουν όμω και πάρα πολλοί επιστημονικοί ενδιασμοί και δαπανούμε δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων ευρώ. Ξέρετε τι λένε οι Αμερικάνοι σε σχέση με αυτό, ότι το ΙΤΕΡ θα στοιχήσει 65 δισεκατομμύρια ευρώ. Εγώ ανησυχώ όμως πάρα πολύ και πραγματικά θα πρέπει να μας πει και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αν υπάρχει για το σύνολο του έργου ένας δημοσιονομικός έλεγχος. Δεν μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε να δίνουμε δισεκατομμύρια ευρώ επαόριστον Α μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για σημαντικέ προκλήσει, όπω ο μετριασμό τη κλιματική αλλαγή. Κυρία Πρόεδρε, χρειαζόμαστε μια πραγματική επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη και από τι Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά και από άλλε χώρε, που θα μπορούσαν πραγματικά να μα πούνε αν μπορεί να πραγματοποιηθεί το σχέδιο αυτό. Και όσον αφορά το υδρογόνο, πολύ ωραία. Έχει γίνει όμω και μία μελέτη που δείχνει ότι χρησιμοποιούμε την ηλεκτρόλυση και δεν ξέρω αν θα πρέπει εδώ πέρα να χρησιμοποιήσουμε και διαφορετικές μεθόδους για την παραγωγή υδρογόνου και το πρόβλημα έπειτα είναι η αποθήκευση. Αυτό είναι η βασική πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε με το υδρογόνο. Εγώ συμφωνώ με αυτά που υπόθηκαν σε σχέση με τον ορίζοντα 2020. Όντω μπορούμε να έχουμε εδώ πέρα μια προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη, αλλά θα αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και τα εμπόδια τα οποία έχουν εντοπιστεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κούς, παραλίγο να σας ξεχάσω. Αλλά να είστε σύντομος παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν έχω στην ουσία ερωτήσεις. Ε, κατανοώ αυτά που ρώτησε η συνάδελφος. Ε, συμφωνώ και εγώ έχω μεγάλες αμφιβολίες για το αν ε, ισχύουν όλα αυτά, αλλά υπάρχουν και διάφορα υποπροϊόντα, διάφορες, ε, διάφορετι, διάφορες ιστορίες, όπως ε, το τεφλόν, ας πούμε, που ήταν παράγω του προγράμματος Απόλλων. Δεν ξέρω βέβαια αν ε, κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο υποπροϊόν θα αξίζει επένδυση 65 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα οικονομικά, εκεί κάτι ξέρω, κάτι κατέχω, βλέπω λοιπόν ότι στις κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου υπάρχει οικονομική επιβάρυνση 179 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή μια σημαντική ε, αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Εσείς πώς το εξηγείτε αυτό, πώς το αιτιολογείτε, διότι δεν αποκόμισα την εντύπωση ότι έχετε καταφέρει και πάρα πολλά θετικά πράγματα με το υδρογόνο. Ισχύει δηλαδή το ότι όσο λιγότερα χρήματα παίρνετε από εμά, τόσο πιο αποτελεσματικοί είστε, διότι σε αυτή την περίπτωση να σα την κόψουμε τη χρηματοδότηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι ιδιαίτερη η λογική που ακολουθείτε. Ωραία, θα δώσω λοιπόν το λόγο στους εκπροσώπους των κοινών επιχειρήσεων και να σας παρακαλέσω μέσα σε τέσσερα λεπτά να έχετε ολοκληρώσει την τοποθέτησή σας. Ας μην εστιάσουμε σε υπερβολικά τεχνολογικά θέματα, δεν είναι ανάγκη να το κάνουμε εδώ. Εμείς είμαστε εδώ για θέματα προϋπολογισμού. Έχετε λοιπόν το λόγο. Ποιος θα ξεκινήσει, κύριε Κάιν. Νομίζω πως δεν χρειάζομαι καν τέσσερα λεπτά, διότι αν κατάλαβα καλά, δύο κύρια ζητήματα υπήρχαν σχετικά με τους καθαρούς ουρανούς. Πρώτον, ε, ο βαθμός, ε, τα ποσοστά εκτέλεξη, 43% το 2018 και ε, τώρα βρισκόμαστε κοντά στο 65%, στο, στα δύο τρίτα δηλαδή. Νομίζω πως ε, όλα βαίνουν καλό σε σχέση με τις απαιτήσει του προγράμματος για το σχέδιο ανάπτυξης. Το σχέδιο ανάπτυξης ε, μάλιστα δημιουργήθηκε στην αρχή του προγράμματος. Και το δεύτερο θέμα ήταν ε, σχετικά με τις συνεισφορές σε είδος. Και εδώ αναφέραμε ότι βρισκόμαστε σε ένα ποσοστό μόχλευσης 2,4%, το οποίο δεν θα είναι φυσικά το τελικό ποσοστό, το οποίο είναι 1,98%. Βρισκόμαστε βέβαια σε καλό δρόμο για να πιάσουμε αυτά τα ποσοστά. Αυτά, αν θυμάμαι καλά. Παρακαλώ, ο επόμενος. Κάποιες ερωτήσεις. Πόσοι εργάζονται για την απαλλαγή και το κόστος. Ένας εργάζεται. Άρα μια χαρά. Γιατί είναι και ιδιαίτερα έμπειροι οι συνεργάτες μας, πρέπει να το τονίσω και αυτό. Έχουμε μόνο 27 άτομα. Άρα μόνο 3% του προϋπολογισμού μας πάει σε διοικητικό κόστος, ενώ θα μπορούσε να ανέβει μέχρι το 5%. Άρα τα πάμε πολύ καλά. Εκτέλεση στον ορίζοντα 20%, 84% μέχρι τέλος του χρόνου, μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε 84% από τους πόρους του ορίζοντα 2020. Πολύ καλό ποσοστό. Οι συμπληρωματικέ δραστηριότητες. Επιτύχαμε το στόχο που έθεσε το Κοινοβούλιο πριν από δύο χρόνια. Τον υπερεύημεν, μάλιστα. Μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς, μάλλον θα έχουμε διπλασιάσει αυτά που μας είχαν ζήτηθει. Αυτό δείχνει ότι ο κλάδος ενδιαφέρεται να επενδύσει σε αυτές τις τεχνολογίες. Η άλλη ερώτηση. Για τη χρηματοδότηση. Τώρα δεν ξέρω αν την κατάλαβα. Από το 2014 που ξεκινήσαμε έχουμε σαφές πρόγραμμα για το πόσα θα επενδύσουμε κάθε χρόνο. Θέλαμε να επενδύσουμε λίγο περισσότερο στην αρχή από ότι στο τέλος. Γι' αυτό είναι έτσι η κατάσταση, γιατί θέλαμε να ξεκινήσουμε με φόρα. Τώρα για τι τεχνικέ ερωτήσει δεν ξέρω τώρα αν έχει έννοια. Θέλετε να απαντήσω για την παραγωγή υδρογόνων. Είναι σαφές. Πρέπει να μην γίνεται μέσω χρήση ορυκτών καυσίμων. Να είναι σαφές. Πρέπει να επιτύχουμε του στόχου των Παρισίων. Και χωρί πυρηνική. Μα δεν έχουμε πυρηνική. Δεν έχουμε πυρηνική ενέργεια. Δεν χρησιμοποιούμε πυρηνική ενέργεια. Εμεί δουλεύουμε μόνο με ανανεώσιμε για την αποθήκευση. Δεν υπάρχει πρόβλημα με την αποθήκευση. Μπορούμε να αποθηκεύσουμε σε κενά πεδία φυσικού αερίου ή σε κατάλληλες σπηλιές. Τεχνικά γίνεται. Το κόστος είναι το θέμα. Γιατί σήμερα δεν υπάρχει τίμημα για την αποθήκευση της, ε, του υδρογόνου. Ξέρετε εάν το δεσμεύσει το υδρογόνο το καλοκαίρι, πρέπει να το χρησιμοποιήσει το χειμώνα. Και ποιο θα πληρώσει την αποθήκευσή του μέχρι τότε. Εδώ είναι το θέμα. Πρέπει να δούμε το χρηματοδοτικό σχήμα. Αυτό δεν ισχύει μόνο για το υδρογόνο όμω, ισχύει για του συσσωρευτέ, για πολλά θέματα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο ή πρόεδρο. Ευχαριστώ για τι ε, τεχνικέ σα ε, απαντήσει. Τώρα και ο εκπρόσωπος Twitter που θα πρέπει να δώσει τεχνικές απαντήσεις και εκείνους. Ναι, ναι, μα μ' αρέσουν τεχνικές απαντήσεις. Για το κεφάλαιο 3 λοιπόν, απαντώντας στις ερωτήσεις του συγκητή, ναι, έχει αλλάξει ο προπολογισμό μας, ο προϋπολογισμός μας και ο προγραμματισμός μας από το 2015. Ο νέος προϋπολογισμός και το αίτημα για την ε, χρηματοδότησή μας έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο. Ο νέος προϋπολογισμός εκπονήθηκε με βάση και τα διδάγματα του παρελθόντος. Γι' αυτό έχουμε τόση αυτοπεποίθηση και θεωρούμε ότι δεν θα τον υπερβούμε τώρα. Και έτσι απαντάω και στο σημείο 10. Ναι, υπήρξαν κάποια προβλήματα, ιδιαίτερα όσον αφορά τις πληρωμές. Όμως ε, έχουμε λοιπόν έναυσμα για να δημιουργήσουμε ένα νέο πιο αποτελεσματικό σύστημα το οποίο επένεσε και το ηλεκτρικό συνέδριο. Έχουμε επαγγελματικού συμβούλους για τα θέματα αυτά. Έτσι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο προγραμματισμό των πληρωμών. Από τότε που είχαμε αυτά τα επεισόδια το 2017 αποδείξαμε ότι μπορούμε να είμαστε πολύ πιο ακριβείς και όριμοι. Και τέλος, υπάρχουν κάποια θέματα επικοινωνίας όσον αφορά την κατάργηση μετά το 2040 την, ε, την πάυση λειτουργίας κάποιων εγκαταστάσεων. Τα λαμβάνουμε υπόψη όλα αυτά που είναι βεβαίως πολύ μακροπρόθεσμα αλλά τα συμπεριλαμβάνουμε στην υποβολή εκθέσεων και τον προγραμματισμό μας. Τώρα για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ερώτηση της κυρίας Ριβαζή. Μα τι είναι αυτό το ίτερ. Είναι έρευνα ή είναι παραγωγή ενέργειας. Και αν δικαιολογούνται οι πόροι που του αποδίδονται, η έρευνα όπως είπα. Το πλάσμα είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα αντικείμενα στο σύμπαν και δεν καταλαβαίνουμε πλήρως ε, πώς λειτουργεί. Και στο ΣΕΡΝ ασχολούμεθα με αυτό, όπου η Ευρώπη δαπανά τόσα και περισσότερα από όσα δαπανά για μας, για να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι καλό να καταλαβαίνουμε το σύμπαν, και νομίζω ότι και αν ακόμη όλα αυτά δεν θα κατέληγαν σε παραγωγή ενέργειας, μόνο ως έρευνα για το πλάσμα θα ήταν αιτιολογημένη η προσπάθειά μας αυτή για το ίτερ. Και αν δείτε ποιο θα μπορούσε να το αποτέλεσμα, δεν είναι υπερβολικές οι δαπάνες. Και πώς όλα αυτά θα συμβάλλουν στο ενεργειακό μείγμα. Δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, είναι σαφές, πριν το 2050. Τι θα γίνει μετά, και αν θα χρειαστούμε τουλάχιστον μία βάση ενέργειας καθαρή και αν μπορούμε να αντικαταστήσουμε την σχάση με τη σύνδεξη, γιατί η σχάση προκαλεί πολλά προβλήματα και έχει πολλά απόβλητα. Γι' αυτό πρέπει να στραφούμε προς άλλα πράγματα, αλλά διάφορα, όχι μόνο προς τη σύνδεξη, αλλά θα μπορούσε να είναι ένα στοιχείο. Και ίσως η σύνδεξη μας επιτρέψει να κλείσουμε όλους τους σταθμούς χάσης. Ξέρετε τι γίνεται στην Ασία, στην Ινδία. Αυτή τη στιγμή δεκάδες πυρηνικοί σταθμοί σχάσης είναι υποκατασκευή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η έρευνά μας μπορεί στο μέλλον να οδηγήσει σε καθαρή και βιώσιμη ενέργεια τουλάχιστον ένα βασικό ποσοστό της. Σας καλώ λοιπόν να επισκεφτείτε το site μας σημάνουν συγγνώμη, όχι εννοώ, όχι το site στο ίντερνετ, να επισκεφτείτε τον, ε, το εργοτάξιό μας να δείτε τι ακριβώς κάνουμε. Ευχαριστώ. Για το Brexit, α, συγγνώμη, ξέχασα για το Brexit. Τα εξής. Πρέπει να το δούμε στο σωστό του πλαίσιο, στη σωστή διάσταση. Είναι μόνο 16% του προπολογισμού μας. Συνεργαζόμεθα πολύ με το ε, Ηνωμένο Βασίλειο. Ξέρετε ότι το μηχάνημα σύνδεξης JET είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο και μας είπαν ότι ενδιαφέρονται στο μέλλον να συνεργαστούν με την ε, Ευρατόμ. Τώρα βέβαια η Επιτροπή θα πρέπει να μας πει αν γίνεται ή δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν είναι δεδεθειμένη να μας πει τώρα, όχι πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια λύση παρόμοια με τη συνεργασία που έχουμε τώρα με την Ελβετία, αλλά είναι νωρί ακόμη για να πούμε τι θα γίνει, γιατί είναι υποδιαπραγμάτευση το θέμα αυτό. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Και ένα λεπτό τώρα για τον εισηγητή, για να ολοκληρώσει. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση. Και θα ήθελα να σας πω ότι ε, στα επόμενα στάδια θα πρέπει να εξετάσουμε στις 20 και 21 Ιανουαρίου του 2020 το σχέδιο έκθεσης σε σχέση με την απαλλαγή αυτή, ενώ στις 29 Ιανουαρίου μέχρι τις 2 το μεσημέρι είναι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης τροπολογίων τα σχέδια εκθέσεων θα εγκριθούν στις 19 και 20 Φεβρουαρίου του 2020 εδώ στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και τους διευθυντές των κοινών αυτών επιχειρήσεων και τους φίλους και τους συναδέλφους της Επιτροπής μας για τις πολύ καλές ερωτήσεις τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε και εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλους τους παρεμβαίνοντες για τη συνεισφορά τους και όλους όσοι συμμετείχαν στη συζήτηση. Ας περάσουμε ευθύ αμέσως στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Περνάμε έτσι στην απαλλαγή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. Please. Σας παρακαλώ πολύ για όσους αποχωρούν από την αίθουσα μην κάνετε θόρυβο. Ε, πολύ ωραία. Λοιπόν, όπως σας είπα, περνάμε στο επόμενο σημείο της σημερινή διάταξη. στο σημείο 5, ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στην αφορά την απαλλαγή για το οικονομικό έτος του 2018 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ πολύ μη θορυβείτε. Yes, please. To move in silence, please. Λοιπόν, μην κάνετε θόρυβος παρακαλώ πολύ. Ας περάσουμε στο επόμενο σημείο της μερίσιας διάταξης, λοιπόν. Για μία ακόμα φορά, σα σας λέω ότι περνάμε στο επόμενο σημείο της μερίσιας διάταξης, ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, απαλλαγή 2018 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους. Να δώσω αμέσως το λόγο στην, στο, στην εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνδεδρίου, την κυρία Ιβάνοβα, για να μας κάνει τη σχετική παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Είναι πάντα για μένα μια ευχαρίστηση να βρίσκομαι εδώ στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού για να σας παρουσιάσω δύο ειδικέ εκθέσεις αυτή τη φορά. Καμία από τις δύο βέβαια δεν έχει συνταχθεί από μένα αλλά ως επικεφαλής του αρμοδίου τμήματος εκπροσωπώ και τους συναδέλφους που δεν μπορούν να είναι σήμερα παρόντες. Ο κύριος Πούφαν που ήταν ο εισηγητής ολοκλήρωσε την θητεία του στο Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, επομένω τον αντικαθιστώ εγώ σήμερα. Όσον αφορά λοιπόν το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους. Εδώ πέρα το σπέρασμά μα είναι ότι η στήριξή του είναι πολύτιμη, αλλά η συμβολή του στη μείωση τη φτώχεια δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους βρίσκεται ακόμα, κινδυνεύει μάλλον από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η καταπολέμηση λοιπόν του κοινωνικού αποκλεισμού και η καταπολέμηση της φτώχειας βρίσκεται στην στρατηγική 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 20 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να βγουν από τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού μέχρι το 2020 σε σχέση με το 2008 και βέβαια αυτό αφορά όλου ιδιαίτερου κάποιες ευάλωτε ομάδες όπως οι νέοι, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι. 3,8 δισεκατομμύρια δίνονται για, από το 2014 και μετά στο ΦΕΑΝΤ, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, με ιδιαίτερη έμφαση στην ακραία φτώχεια και την αντιμετώπιση της φτώχειας των, των νέων, των παιδιών της καλύτερης πρόσβασης σε τρόφιμα και της καλύτερης πρόσβασης σε στέγαση. Το Ταμείο αυτό Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους έχει επιφέρει τρεις βασικές αλλαγές. Έχουμε ηλική συνδρομή, καθώς επίσης και μέτρα κοινωνικής ένταξης. Τα κράτη-μέλη μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο επιχειρησιακά προγράμματα εντελώς διακριτά και περάσαμε από την DG Agri στην DG Employment όσον αφορά δηλαδή την επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπετε τα τρία βασικά ερωτήματα τα οποία θέσαμε. Δεν πρόκειται να σας τα διαβάσω, τα βλέπετε στη διαφάνεια. Πρόκειται ουσιαστικά για τις τρεις βασικές διερευνητικές γραμμές που ακολουθήσαμε στο πλαίσιο της έκθεσης ελέγχου και θα σας δώσω με τις επόμενες διαφάνειες κάποιες περαιτέρω λεπτομέρειες. Βλέπετε ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να επιλέξουν, όπως σας είπα, δύο ξεχωριστά επιχειρησιακά προγράμματα, να εφαρμόσουν ακόμα και τα δύο, αλλά κανένα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επέλεξαν και τα δύο. Περιορίστηκαν είτε στο ένα είτε στο άλλο. Και είδαμε ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη τελικά επέλεξαν το πρώτο επιχειρησιακό πρόγραμμα που είχε να κάνει με την επιστητιστική βοήθεια και την τεχνική συνδρομή μαζί με κάποια συνοδευτικά μέτρα. Το δεύτερο όμως επιχειρησιακό πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει ηλική συνδρομή, επιστηστική βοήθεια, αλλά κυρίως μέτρα κοινωνικής ένταξης που απευθύνονται στους πλέον απόρους, στις πιο μειονεκτούσες ομάδες. 24 κράτη-μέλη επέλεξαν το πρώτο επιχειρησιακό πρόγραμμα, 10 μόνο δίνουν επιστηστική βοήθεια και ένα ηλική συνδρομή μόνο. Τα υπόλοιπα κράτη-μέλη παρέχουν και τα δύο, δηλαδή και επιστηστική βοήθεια και ηλική συνδρομή. Και εν γέννη το συμπέρασμά μα είναι ότι το πρώτο επιχειρησιακό πρόγραμμα αντιστοιχεί περίπου στο 97,8% του συνολικού προπολογισμού του Ταμείου Ευρωπαϊκή Βοήθεια προ του Απόρου. Στο πρώτο αυτό επιχειρησιακό πρόγραμμα, η επιστηστική βοήθεια είναι το 84% του προπολογισμού και βάσει των δεδομένων αυτών μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η βασική βοήθεια ήταν κυρίω επισητιστική συνδρομή μέσω του πρώτου επιχειρησιακού προγράμματο. Και τέσσερα, όπω σα είπα, μόνο κράτη-μέλη, η Γερμανία, η Δανία, οι κάτω χώρε και η Σουηδία, επέλεξαν το δεύτερο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Κάνω όμω και μία έρευνα που απευθυνόταν και στις 28 διαχειριστικές αρχές, 23 απάντησαν, λέγοντάς μας ότι το φεάτι ήταν πολύ σημαντικό ή έστω σημαντικό για την υποστήριξη προς τους πιο απόρους και η λεκτική μας ομάδα πήγε και σε κάποια σεμινάρια του δικτύου της ΦΕΑΤ που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκεί πραγματικά μπορούσαμε να καταλάβουμε τη σημασία της υποστήριξης από το ΦΕΑΤ για εκκλησίες, για κοινωνικές πρωτοβουλίες, για μη κυβερνητικέ οργανώσεις που προσπαθούν να βοηθήσουν τους απόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά η σημασία του ΦΕΑΤ στο γενικότερο πλαίσιο σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο δεν είναι ακόμα πάρα πολύ γνωστή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ως προς αυτό δεδομένα, προκειμένου να μπορούμε πραγματικά να συγκρίνουμε τη μία χώρα με την άλλη. Δεν υφίστανται αυτά τα διαστοριακά δεδομένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την πτυχή της φτώχεια. Τα νέα στοιχεία των συνοδευτικών μέτρων στα πλαίσια του πρώτου επιχειρησιακού προγράμματος έχουν ως στόχο να υπάρχει μια πιο στοχευμένη προσέγγιση για την κοινωνική ένταξη και βέβαια χαιρετίζουμε τα μέτρα αυτά γιατί καθιστούν σαφή βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα. Τα περισσότερα κράτη-μέλη στα οποία κάναμε έρευνα δεν μπορούσαν να μας πούνε το μερίδιο στο οποίο αντιστοιχεί το ΦΕΑΤ όσον αφορά το στέλνο του προπολογισμού που δίνουν για την υποστήριξη προς τους απόρους. Βλέπετε πάντως ότι μπορέσαμε να έχουμε κάποιες εκτιμήσεις για κάποιες χώρες και εδώ πραγματικά μπορούμε να εντοπίσουμε τη γενικότερη σημασία του ΦΕΑΤ που μπορεί να φτάσει ακόμα και το 60% σε κάποιες χώρες όπως βλέπουμε. Τώρα, η στόχευση, η στοχοθέτηση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό προκειμένου τα, τα ευρωπαϊκά αυτά ταμεία να έχουν ένα πραγματικό επιτόπου αποτέλεσμα, ένα ίμιση μόνο των κρατών μελών που ελέγχθηκαν πραγματικά έχουν εντοπίσει συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες που μπορούν να επωφεληθούν από τα επιχειρησιακά προγράμματα. Οι περισσότερες χώρες ορίζουν τους απόρους με ένα πολύ ευρύ και γενικό τρόπο και ουσιαστικά προσπαθούν μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων να συνεχίσουν το παλαιότερο πρόγραμμα επισητιστικής βοήθειας. Το ίμιση των κρατών μελών συνδυάζουν την βοήθεια από το ΦΕΑΤ με άλλα κοινωνικά μέτρα τα οποία δίνονται από το κράτος μέλος και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούν με ένα πιο αυστηρό τρόπο να παράσχουν βοήθεια προς τους απόρους. Όσον αφορά τα συνοδευτικά μέτρα είναι πολύ σημαντικά καθότι η επιστημική βοήθεια από μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα βαθύτερα αίτια της φτώχειας. Όπως βλέπουμε στην διάμεση αξιολόγηση το ΦΕΑΤ είναι ένα πρόγραμμα για τους ανθρώπους, για την υποστήριξη των πολιτών και όχι απλώς ένα πρόγραμμα διανομής τροφίμων. Τα συνοδευτικά μέτρα που επιλέγουν τα κράτη-μέλη διαφέρουν πολύ από το ένα στο άλλο και είναι δύσκολο να κάνουμε τώρα μια σύγκριση. Έχουμε διάφορες πληροφορίες που δίνονται από κάποια φυλάδια που απευθύνονται κυρίω στου αστέγους για το πού μπορούν να βρουν στέγαση. Έχουμε σε κάποιες άλλες χώρες πιο εξατομικευμένα προγραμμά, προγράμματα στήριξης. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμα κοινού δείκτες όσον αφορά τα συνοδευτικά μέτρα, ούτε δείκτες μέτρησης των αποτελεσμάτων των μέτρων αυτών. Αναγνωρίζουμε πάντως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στα κράτη-μέλη όσον αφορά τα συνοδευτικά μέτρα. Πάντω, τα επιχειρησιακά προγράμματα και τα δύο θα πρέπει να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο, προκειμένου να αλληλοσυμπληρώνονται καλύτερα με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τα σχετικά του μέτρα. Τώρα, όσον αφορά τι συστάσει του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τρεις είναι οι βασικές μα συστάσει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και προς τα κράτη-μέλη. Πρώτον, όταν εγκρίνονται επιχειρησιακά προγράμματα στα πλαίσια του νέου ESF+, θα πρέπει να απαιτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνουν τα κράτη-μέλη μια καλύτερη στόχευση της βασικής επιστημιστική και ηλικής βοήθειας προς αυτούς που την έχουν περισσότερο ανάγκη, περιγράφοντας καλύτερα την κατάσταση της φτώχειας, εντοπίζοντας καλύτερα τις μειονεκτούσες ομάδες και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για να φτάσει σε αυτούς η βοήθεια. Και θα πρέπει επίση επίσης να έχουμε καλύτερα σημεία αναφοράς, δείκτες αναφοράς, ποσοτικοποιημένους δείκτες. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε την παροχή μέτρων κοινωνικής ένταξης για τους δικαιούχους της βασικής ηλικής συνδρομής υπό το νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus για την περίοδο 2021-2027 Επίσης, είναι σημαντικό μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων φορέων να έχουμε καλύτερη επαφή με τους πλέον απόρους. Αυτό θα πρέπει να τηρηθεί στο πλαίσιο του νέου ΦΕΑΔ. Τα κράτη-μέλη τα οποία θα χρησιμοποιήσουν τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να παρέχουν επιστηστική βοήθεια ή άλλη τεχνητή ηλική συνδρομή μάλλον, θα πρέπει να περιλαμβάνουν και συνοδευτικά μέτρα, τα οποία θα συμπληρώνουν τη βασική επιστημιστική ή ηλική βοήθεια ή θα πρέπει να εντοπίσουν τα επιχειρησιακά εκείνα προγράμματα, τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν συνοδευτικά μέτρα προς τους δικαιούχους. Η τρίτη μας σύσταση έχει να κάνει με την βελτίωση της αξιολόγησης όσον αφορά την κοινωνική ένταξη που παρέχει το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους όσον αφορά πάντα τους τελικούς δικαιούχους. Αυτά κυρία Πρόεδρε, ας μην αναλώσω περισσότερο χρόνο. Είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήσει ή παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Ιβάνοβα για την παρουσίαση σας αυτή. Να δώσω το λόγο στην κυρία Γκραπίνη τώρα που είναι η συγγήτριά μας. Έχετε κι εσείς μέγιστο 10 λεπτά κυρία Γκραπίνη. Vreau să, de la bun început, să salut raportul special al Curții de Conturi σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίζω και εγώ την έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου για το Ταμείο και να ευχαριστήσω την κυρία Ιβανόβα για την παρουσίαση της έκθεσης. καθώς και για τις παρατηρήσεις και συστάσεις που έγιναν. Είναι πολύ σημαντικές για εμάς γιατί βλέπουμε τις φελτιώσεις στην διαδικασία αυτή. Η κυρία Ιβανόβα ανέφερε ότι ακόμα και αν το ταμείο αυτό χρησιμοποιείται στο πλαίσιο μιας ε, Ευρώπης ευημερίας, πάρα πολλοί πολίτες ε, είναι αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της φτώχειας. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εξετάσει τις δυνατότητες ε, που μπορεί να χρησιμοποιήσει έτσι ώστε να έχει το μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο το ταμείο αυτό. Μας είπατε ότι πρέπει να βγάλουμε εκατομμύρια ανθρώπων από τη φτώχεια μέχρι το 2020. Εγώ νομίζω ότι χρειάζονται δραστικά μέτρα. Και η συζήτηση αυτή έρχεται στην κατάλληλη στιγμή, διότι μας δίνει μια γενικότερη εικόνα του τι συμβαίνει γύρω μας. Όμως το ελεκτικό συνέδριο θεωρεί ότι μας είπε μάλλον ότι το πρόγραμμα αυτό είναι περισσότερο επισητιστικό. Δεν νομίζω ότι στο μέλλον θα πρέπει να περιοριζόμαστε στον επισητιστικό τομέα, αλλά να καταπολεμήσουμε τα αίτια του προβλήματος. Και γι' αυτό χρειάζεται να σκεφτούμε μακροπρόθεσμα. Το ελεκτικό συνέδριο δεν μπορούσε να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του Ταμείου, διότι μας είπατε κι εσείς οι ίδια ότι τα δεδομένα ήταν ελλειπή, ανεπαρκή. Ε, και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μας πει τι σκοπεύει να κάνει στο μέλλον έτσι ώστε να διορθωθεί αυτό το θέμα της ανεπαρκείας των ε, δεδομένων. Θα μπορούσαμε λοιπόν να το σκεφτούμε, όμως ε, εγώ επιθυμώ να τονίσω ορισμένα στοιχεία. Υπάρχει, είπατε, η δυνατότητα να συνδυαστεί η επιστημιστική βοήθεια με διάφορα μέτρα καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Νομίζω πως γνωρίζουμε όλοι εδώ πώ υπάρχουν ε, κράτη-μέλη τα οποία παρότι είναι αρκετά ανεπτυγμένα αντιμετωπίζουν προβλήματα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Και νομίζω θα συμφωνήσετε ότι ο κατάλληλος έλεγχος των ε, αποτελεσμάτων μαζί με τα συνοδευτικά μέτρα ε, που αναφερθήκατε και εσείς σε αυτήν την ε, λογική της παρέμβασης ε, θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση των μέτρων αυτών. Μας είπατε κι εσείς ότι υπάρχει αναπάρκεια στοιχείων σχετικά με τα μέτρα καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Και έχω συγκεκριμένες ερωτήσεις και για το ελεκτικό συνέδριο και για την Κομισιόν. Πρώτον, θεωρείτε πως είναι πλέον αργά να, για να βελτιωθεί η εφαρμογή του ΦΕΑΔ έτσι ώστε να καταφέρει να ασχοληθεί με τα προβλήματα που εντόπισε το ελεκτικό συνέδριο ή θεωρείτε πως ε, κατά την παρούσα περίοδο μπορούν να γίνουν κινήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Οι αδυναμίες επίσης που εντόπισε το ελεκτικό συνέδριο έχουν να κάνουν με την υφιστάμενη νομοθεσία ή υπάρχουν άλλα αίτια. Διότι αυτό πρέπει να το δούμε. Αν είναι πρόβλημα νομοθετικού πλαισίου, μπορούμε να παρέμβουμε και οφείλουμε να παρέμβουμε. Το ηλεκτρικό Συνέδριο συμφώνησε σχετικά με ε, την σύσταση 1 παράγραφο σε για τους ποσοτικούς στόχους, δηλαδή τι λύσεις ε, μπορούμε να φανταστούμε έτσι ώστε να βελτιωθεί η εποπτεία της ε, χρήσης του Ταμείου για τους απόρους με τις διάφορες πτυχές του και παράδειγμα εθελοντική εργασία και με προϋπόθεση τον σεβασμό της αξιοπρέπειας των τελικών δικαιούχων πάντα συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Και ερώτηση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μπορούσατε να μας δώσετε συγκεκριμένα παραδείγματα χρήσης του Ταμείου με χρήσης του Ταμείου όπου θα ληφθούν υπόψη οι συστάσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου. Θα ήθελα λοιπόν να ολοκληρώσω λέγοντας ότι ένας ε, σημαντικός ε, στόχος που θα πρέπει να έχουμε και εμείς και το Συμβούλιο είναι να εξασφαλίσουμε μία ομοιογενή ανάπτυξη στην Ευρώπη έτσι ώστε να βγει ο κόσμος από τη φτώχεια, να μην υπάρχουν απομονωμένες, αποκλεισμένες περιοχές όπως δηλαδή κατέληξε και το ελεκτικό συνέδριο, το ΦΕΑΤ θα πρέπει να είναι ένα μέσο που θα παρέχει επισκεπτική βοήθεια και γενικότερη στήριξη σε όσους έχουν ανάγκη, αλλά θα πρέπει να συντονιστεί και με άλλους τομείς πολιτικής, όπως την υγειονομική περίθαλψη, την παιδεία για παράδειγμα, αλλά και με ιδιωτικές πρωτοβουλίες, δημόσιου δημόσιο-ιδιωτικού τομέα και άλλα. Το ΦΕΑΤ είναι μια καλή ιδέα, χρειάζεται όμως καλύτερη εποπτεία, καλύτερο έλεγχο και συγχρονισμένη δουλειά μαζί με τα κράτη-μέλη, διότι ο στόχος μας είναι ακριβώς αυτοί που έχουν περισσότερη ανάγκη. Να ευχαριστήσω λοιπόν το ελεκτικό συνέδριο που ήρθε και τους ε, εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρώ πως θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε συγκεκριμένες απαντήσεις για να αναπτύξουμε συγκεκριμένα μέτρα. Σας ευχαριστούμε κυρία Γκραπίνη. Ο κύριος Χριστοφόρου τώρα έχει το λόγο που είναι και Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, είναι σημαντική συζήτηση που γίνεται σήμερα γιατί είναι σημαντικότατο το θέμα που συζητάμε όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκύπτει σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εξάλληψη της φτώχειας. Θέλω να εξάρω πραγματικά την, ε, το μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, την κυρία Ιβάνοβα, για τις εύστοχες παρατηρήσεις και εισηγήσεις της, καθώς και την ε, αγαπητή συνάδελφον εισηγήτρια, με την οποία συμφωνώ απόλυτα, και βρίσκουμε στην ίδια γραμμή και στην ίδια πορεία πλεύσης όσον αφορά την αντιμετώπιση και τη διαχείριση αυτών των ζητημάτων που άπτονται με τη διαχείριση τη φτώχεια και του περιορισμού του κοινωνικού αποκλεισμού μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ω κοιόδης εισηγητής πραγματικά θεωρώ ότι ο στόχο όλων μα θα έπρεπε να είναι αυτό το ταμείο να έχει ένα και μοναδικό στόχο. Κανένα Ευρωπαίο πολίτη να μην κινδυνεύει από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό κανένας Ευρωπαίος πολίτης να μην είναι επέτης, κανένας Ευρωπαίος πολίτης να μην είναι άστεγος. Εάν πραγματικά θέλουμε αυτό το ευρωπαϊκό οικοδόμημα να το αποκαλούμε ως οικοδόμημα πολιτισμού, ως οικοδόμημα πρόοδου και ευημερία, αυτό που συμβαίνει με την καταγεγραμμένη σε υψηλά ποσοστά φτώχεια αποτελεί πραγματικά προσβολή και ντροπή για όλους μας. Το ότι διατίθενται 3,8 δισεκατομμύρια είναι ένα σημαντικό ποσό και δεν το μηδενίζουμε, όπω δεν μηδενίζουμε και τι κοινωνικέ πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ανήκουμε σε αυτού που λένε ότι η Ευρώπη δεν κάνει τίποτα κοινωνικό και δεν έχει κοινωνική ευαισθησία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κοινωνική ευαισθησία και το αποδεικνύει και με αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο που είναι καθαρά κοινωνικό και έχει να κάνει με του άπορου. Αλλά για να μπορέσουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο τη φτώχεια που φαίνεται ότι δεν αντιμετωπίστηκε μέχρι σήμερα, πρέπει να πάρουμε μια σημαντική απόφαση που έχει να κάνει με τον προπολογισμό επειδή ανήκω στην Επιτροπή Προπολογισμού, θέλω να πω ότι είμαι θειασότη του να αυξηθεί η συνεισφορά των χωρών μέλο του 1,3%. Και μαζί με την αύξηση αυτή του 1,3% πρέπει να δεσμεύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, να δεσμεύσουμε τον προπολογισμό, το 1% των χρημάτων του προπολογισμού να πηγαίνουν για την αντιμετώπιση τη στόχια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Όσε επιτυχίε και να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, Εάν δεν κατορθώσει να περιορίσει τα ποσοστά φτώχεια και κοινωνικού αποκλεισμού, δεν μπορεί να λογίζονται επιτυχίε. Άρα, επιτυχία για μα θα είναι όταν θα εξαλειφθεί πλήρω η φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με αυτόν τον τρόπο θα είναι και η καλύτερη διαφήμιση για την επιτυχία του ευρωπαϊκού μοντέλου. Στην πατρίδα μου, την Κύπρο, εφαρμόζεται ένα ισχυρό μέτρο για την αντιμετώπιση τη φτώχεια και του κοινωνικού αποκλεισμού σε περίοδο οικονομικής κρίσης πριν πέντε χρόνια όταν η Κύπρος βρισκόταν στα όρια της χροκοπίας η κυβέρνηση τότε πήρε την γενναία απόφαση να εφαρμόσει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που για μονήρι άτομα αγγίζει τα 600 με 700 ευρώ μηνιαίως και για οικογένειες υπερβαίνει τα 1000-1200 ευρώ ένα σημαντικό ένασμα για την πραγματική αντιμετώπιση τη φτώχεια και περιορισμών του κοινωνικού αποκλεισμού. Και ήθελα να ξέρω αν χώρε που παίρνουν μόνε του αυτέ τι πρωτοβουλίε, όπω η Κύπρο και πιθανώ και άλλε, αυτή είναι η αποστολή του Ταμείου, να συνεπικουρήσει αυτέ τι χώρε για να αναλάβουν και οι χώρε μερίδιο τη ευθύνη και του κόστου για να αντιμετωπιστεί αυτό ε, το πραγματικά νοσηρό κοινωνικό φαινόμενο που όπως είπα προσβάλλει και δεν τιμά κανένα από όλους μας. Άρα θεωρώ πολύ σημαντικό εάν εφαρμοστεί το ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα εκ των πραγμάτων δεν θα υπάρχει Ευρωπαίος πολίτης που θα είναι κάτω από το όριο της στόχιας θα κινδυνεύει με κοινωνικό αποκλεισμό και η συνεργασία των χωρών μελών με τον προπολογισμό των δικών μας και με τις πολύ σημαντικές συζητήσεις τόσο του ελεκτικού συνεδρίου όσον και της αγαπητής συναδέλφου εισηγήτριας πιστεύω ότι θα πετύχουμε το στόχο μας που δεν είναι τίποτα άλλο, είναι κοινός στόχος για να μην υπάρχει Ευρωπαίος πολίτης που θα κινείται μέσα σε αυτά τα ιδιαίτερα τροπιαστικά κοινωνικά ε, πλαίσια που είναι του κοινωνικού αποκλεισμού, τη στόχιας και της εξαθλίωσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ κύριε Χριστοφόρου για την παρέμβασή σας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις από τους άλλους παρευρισκόμενους συναδέλφους. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Μα πάντα μου άρεσε η εξή έκφραση. Αν δώσεις ε, στον ψαρά ένα ψάρι θα έχει να φάει μια μέρα. Μάθε του να ψαρεύει θα μπορεί να θρέψει για πάντα την οικογένειά του. Και άμα του μάθεις πώς να φτιάχνει και το καλάμι του και την καθετή του, τότε θα μπορέσει να τραφεί και όλο το χωριό, όταν μιλάμε για φτώχεια. Να μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά είναι μια διαδικασία. Δεν βοηθάει πολύ να μοιράζουμε λεφτά. Πρέπει να δώσουμε τις ικανότητες ε, στους συμπολίτες μας να πάρουν ε, το πεπρωμένο τους στα χέρια τους, να εξαλειφθεί η φτώχεια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό όταν συζητάμε τέτοια θέματα. Οι πόροι πρέπει να αξιοποιούνται ούτω ώστε να αποκτήσουν οι άνθρωποι την ικανότητα και την οτροπία να παλέψουν για να βγουν από τη φτώχεια. Ευχαριστώ πολύ. Και εμεί σα ευχαριστούμε. Τώρα το λόγο για ένα λεπτό έχει ο κύριος η κυρία Στρουγκάριο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αντικαθιστώ την συνάδελφο που είναι σκιώδη συζυγήτρια, η οποία, όπως σας είπα, δεν μπορεί να παρευρεθεί εδώ. Παρ' όλα αυτά, παίρνω τον λόγο εκ μέρους της. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την κυρία Ιβάνοβα. Σας ευχαριστώ, λοιπόν, για την ε, παρουσίαση αυτής της ειδική έκθεσης. Συμφωνώ με την εισηγήτρια την κυρία Γκραπίνη και στηρίζω τη θέση της εκ μέρους της ομάδας Renew Europe. Θεωρώ ότι θα πρέπει στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027 να ενθαρρύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, επικεντρώμενοι όμως στις επιδόσεις προκειμένου το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους να συνάδει με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει των συστάσεων και συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου και όσον αφορά θεματική προγραμματική μάλλον περίοδο 2021-2027, μολονότι οι ελεγκτές είπανε ότι το ΦΕΑΝΤ δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να προωθήσουν και να αντιμετωπίσουν μάλλον την, τον κοινωνικό αποκλεισμό και να προωθήσουν την κοινωνική ένταξη, ελάχιστα είναι τα μέτρα, 2,5% μόνο του προπολογισμού ουσιαστικά, που δίνεται στην κοινωνική ένταξη. Και δυστυχώ δεν έχουμε την απαραίτητη παρακολούθηση για τα υπόλοιπα μέτρα γιατί δεν έχουμε ποσοτικού στόχου. Θα ήθελα λοιπόν να μας πει το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνίδρο ποιου μηχανισμούς θα υιοθετήσει προκειμένου να αξιολογεί καλύτερα τις επιτυχίες των κρατών μελών. Αυτή τη στιγμή βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητήσει από τα κράτη-μέλη να εμπλακούν λίγο περισσότερο στα προγράμματα κοινωνική ένταξη. Περαιτέρω προσπάθειε επίση πρέπει να καταβληθούν προκειμένου να γίνει μία μετάβαση από το ΦΕΑΤ προ το ESF. Αν δεν έχουμε όμω αρκετά διαστοριακά δεδομένα αλλά και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μα πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θα κάνει. Ποιε είναι οι συστάσει του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να διαχέονται καλύτερα τα αποτελέσματα του ΦΕΑΝΤΑ σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν και περισσότερα κράτη-μέλη. Και συμφωνώ απόλυτα με την εισηγήτρια ότι η εξάλληψη της φτώχειας ουσιαστικά σημαίνει να ενισχύσουμε και τους πολίτες, δηλαδή να συνδυάσουμε την άμεση επιστηστική βοήθεια με εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς επίσης και με προγράμματα κοινωνικής ένταξης. Και νομίζω ότι για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο θα πρέπει εκεί να επικεντρωθούμε περισσότερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο για πέντε περίπου λεπτά στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην εκπρόσωπο μάλλον, την κυρία Ιβάνκοβιτς Τσένκεβιτς. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία Ιβάνοβα, θα ήθελα καταρχάς ε, να πω πόσο καλωσορίζουμε την έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου και χαιρόμαστε πολύ που το Ελεκτικό Συνέδριο αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία του ΦΕΑΝΤ. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τις διαφορές μεταξύ του ΦΕΑΝΤ και του προηγούμενου προγράμματος. Για μας ε, το ΦΕΑΝΤ είναι το βασικό μέσο στήριξης ε, των απόρων. Παρέχει επισητιστική και ουσιαστική υλική βοήθεια, αλλά και μέτρα καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Και αυτή η στήριξη παρέχεται σε ένα μεγάλο ποσοστό των απόρων, έτσι ώστε να αλλάξει πραγματικά η ζωή τους. Λέμε ότι με βάση τους υπολογισμούς μας, το ΦΕΑΝΤ βοηθά περίπου 30 εκατομμύρια πολίτες μεταξύ 2013 και 2017 και να σας πω εδώ ότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι υπολογισμοί αυτοί έχουν γίνει από διάφορους ε, συνεργαζόμενους οργανισμούς οι οποίοι ασχολούνται με ε, θέματα στήριξης των απόρων. Παρά λοιπόν ε, το περιορισμ, τις περιορισμένες δυνατότητες του ΦΕΑΔ κατάφερε να φτάσει σε 30 εκατομμύρια πολίτες μέσα σε τρία χρόνια και τα στοιχεία που έχουμε για το 2018 το επιβεβαιώνουν. Η μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση που κάναμε έχει επιβεβαιώσει την αποτελεσματικότητα, την ε, συνεκτικότητα και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του ΦΕΑΝΤ. Τώρα για τον επόμενο μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κομισιόν προτείνει να ενσωματωθεί το ΦΕΑΝΤ με τα άλλα χρηματοδοτικά μέσα υπό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ. Ε, θα συμπεριλαμβάνει μέτρα κατά πολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και άλλα κοινωνικά μέτρα που θα ενισχύσουν την ε, διάσταση αυτή. Και η συγγήτρια και οι συνεισηγητές ε, τόνισαν αμφότερη την σημασία που έχουν τα συνοδευτικά μέτρα, διότι στο πεδίο εφαρμογή του υφιστάμενου CSF και του προηγούμενου που ξεκίνησε πριν από περίπου 15 χρόνια, το στοιχείο της κοινωνικής ενσωμάτωσης πάντα ε, αναφερόταν στα προβλήματα αυτά και στην ε, δύσκολη μειονεκτική θέση που έχουν τα άτομα αυτά στην κοινωνία. Και θεωρεί λοιπόν ότι το ΦΕΑΝΤ είναι ένα πρόσθετο ε, βοηθητικό μέσο, ένα πρόσθετο εργαλείο για να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο αυτό. Πάντα σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, τα οποία γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες των πολιτών τους. Αν ε, παρατηρήσουμε τη σύσταση της ε, βοήθειας ε, μέσω του Ταμείου, παρατηρούμε ότι από τα 13 εκατομμύρια πολιτών που επωφελούνται, οι γυναίκες είναι πάνω από τους μισούς, τα παιδιά αποτελούν το 13% ε, των ε, συνολικών δικαιούχων. Μετά, μετανάστες και άλλες ε, μειονότητες επίσης περίπου 13%, οι ηλικιωμένοι ηλικίες πάνω από 65 ετών πάλι 8,9%, άστεγοι 4%. Φτάνουμε σε ένα σύνολο περίπου 60% των τελικών δικαιούχων του Ταμείου. Και αν συγκρίνουμε την ομάδα αυτή με τα μέτρα υπό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που χρησιμοποιούνται από τα κράτη-μέλη, τότε θα δείτε ότι ε, υπάρχει μία συμφωνία σε αυτό. Πιάνει όλα τα ε, όλες τις ε, ομάδες. Το Ταμείο λοιπόν παρέχει επισητιστική και ηλική βοήθεια, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να λειτουργήσουμε καθοδηγητικά και να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις για εκείνους που το έχουν ανάγκη, για τους απόρους, πάντα με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Να επανέλθω λίγο στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ. Υπό το ταμείο λοιπόν αυτό θέλουμε να κρατήσουμε τα πράγματα απλά, να έχουμε ένα απλό πλαίσιο εφαρμογής, επισητιστικής και ηλικής βοήθειας. Μπορεί να το έχετε δει ήδη στα περισσότερα κρατημέλη να εφαρμόζεται ε, κατά αποκοπή ποσά. Αυτό έχει αποδειχθεί μία καλή λύση για την εκτέλεση των ε, project του Ταμείου. Ταυτόχρονα υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις που στοχεύουν στους απόρους που θα υπάρχουν και στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Πλάς. Σας παρακαλώ, λέει η Πρόεδρος, πιο αργά να μιλάτε. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να γνωρίζουμε ότι έχουμε προτείνει μία ελάχιστη ε, κατανομή σε συγκεκριμένα επιχειρησιακά προγράμματα, δηλαδή το 2% των διαθέσιμων πόρων στην επιμερισμένη διαχείριση. Μετά, σε επίπεδο ένωσης στοχεύουμε στο 4%. Να μείνει δηλαδή σταθερή η στήριξη σε σχέση με την ε, περίοδο που διατρέχουμε. Ε, τώρα σε ό,τι αφορά τις συστάσεις, όλες οι συστάσεις για την επόμενη προγραμματική περίοδο για ε, τις ε, νομοθετικές προτάσεις παραμένουν υπό διαπραγμάτευση από τους συνομοθέτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Αγγέλικα έχει μια ερώτηση. Ναι, μια παρατήρηση. Φτώχεια σημαίνει απόγνωση. Χρειάζεται μία ελάχιστη διασφάλιση, βοήθεια. Αλλά δεν βοηθάει την κοινωνική ισότητα. Και το βασικό είναι να υπάρχει εκπαίδευση, να υπάρχει οικονομική δραστηριότητα, να συνεργαζόμεθα με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις. Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε μία μόνιμη καταπολέμηση και εξάλληψη της φτώχειας. Πρόεδρος. Ιλιάνα, Χαιρετίζω την παρουσία σου. Με συγχωρείς που χρειάστηκε να βγω γιατί έπρεπε να τηλεφωνήσω. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Βλέπω δεν έχουμε χρόνο, άρα θα είμαι σύντομη. Ευχαριστώ την κυρία Κραπίνη, την εισηγητριά μας για τη θαυμάσια εργασία της και τις παρατηρήσεις και τους κοιόδης. Συμφωνώ με όλα τα σχόλια που κάνατε. Όντως, η μείωση της φτώχειας είναι βασικό στοιχείο της στρατηγικής ε, για το 2020 και το ΦΕΑΤ θα βοηθήσει να βγάλουμε τουλάχιστον 20 εκατομμύρια συμπολίτε μας από το, τον κίνδυνο φτώχειας. Αλλά δεν μπορεί να λύσει μόνο του το ΦΕΑΤ το πρόβλημα. Μπορεί απλώς να παίξει συλλογματικό ρόλο. Πρέπει να υπάρξουν και άλλες πολιτικές. και είναι ελάχιστο αυτό το 3,8 δι σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες. Είναι προφανές. Με 3,8 δις θα λύσουμε το πρόβλημα της στόχιας. Καλή ιδέα. Είναι, βελτιώνει το προηγούμενο πλαίσιο, αλλά πολλά μπορούν να βελτιωθούν. Και τα λέει η έκθεση. Το βασικό λοιπόν είναι πραγματικά να μάθουμε στους ανθρώπους να ψαρεύουν και να φτιάχνουν και τον ε, κατάλληλο εξοπλισμό. Βεβαίως μας ενδιαφέρει η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, η ένταξη, για να βελτιώσουμε Κοιτάξτε, στόχος του ελέγχου ήταν να δούμε το σχεδιασμό του προγράμματος. Δεν εξετάσαμε την εφαρμογή. Αλλά το έχουμε υπόψη μας. Θέλουμε να δούμε και πόσο αποτελεσματική θα είναι η εφαρμογή, αλλά χρειάζεται χρόνος. Ελπίζουμε να ικανοποιήσει τις προσδοκίες μας. Καθορίζει δύο διαφορετικούς τρόπους με, τον οποίο, με τους οποίους θα μπορούσε να αξιοποιηθεί το ΦΕΑ, είτε μέσω συνέχισή του προγράμματος ε, γευμάτων ή μέσω βελτίωσης της ε, ένταξης. Οι αδυναμίες έχουν να κάνουν με το παρόν νομοθετικό πλαίσιο, από την άλλη μεριά. Το πλαίσιο ήταν διτό, γιατί ήταν αποτέλεσμα συμβιβασμού μεταξύ των κρατών μελών. Πρώτα απ' όλα να συνεχιστεί από τη μία πλευρά η επιστηστική βοήθεια, η παροχή γευμάτων, κάτι που γίνεται εδώ και καιρό, και άλλε δυνατότητε που αναφέρθηκαν επίση, προβλέπονταν, πιο καινοτόμε και δεν καταλήξαμε παρά τα στοιχεία που συλλέξαμε ότι είναι αδύναμη η εφαρμογή του. Να δούμε τελικά πόσο θα είναι αποτελεσματική η εφαρμογή του βέβαια. Το έχουμε υπόψη μας. Και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις θαυμάσιες ε, ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον εισηγητή, του Σκιώδης. Να περάσουμε τώρα στην ειδική έκθεση 2019. Α, με συγχωρείτε αγαπητοί συνάδελφοι. Α, η, και η κυρία Γραπίνη ήθελε το λόγο. Συγγνώμη, πρέπει να φύγω. Λυπάμαι. Αλλά φεύγω πολύ ικανοποιημένη γιατί όλοι οι συνάδελφοι από όλες τις πολιτικές ομάδες τόνισαν ότι είναι πολύ σημαντικό να δράσουμε ούτως ώστε ένα τμήμα του πληθυσμού μας να βγει από τη φτώχεια. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που πήραν το λόγο και ευχαριστώ και την Επιτροπή και το Λεκτικό Συνέδριο για τις απαντήσεις σας και αναμένουμε και δράση γιατί το βλέπουμε και από τη σημερινή συζήτηση μόνη και μόνη η ύπαρξη του Ταμείου δεν τα επιλύει όλα πρέπει να συνδυαστεί η δράση του Ταμείου με άλλες πολιτικές. Και εγώ στη χώρα μου αγωνίζομαι από τότε που εξελέγει, ούτως ώστε να βελτιωθεί η επαγγελματική κατάρτιση, ούτως ώστε οι νέοι μας να μπορέσουν οι ίδιοι να βοηθηθούν, να τους βοηθήσουμε να βοηθηθούν, να αυτοβοηθηθούν. Γιατί ξέρουμε ότι πολλοί δεν έχουν δουλειά γιατί δεν έχουν τις δεξιότητες. Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε και θέσει εργασία όμω, γιατί και άτομα με προσόντα δεν βρίσκουν θέσει εργασία ε, στον ε, τόπο κατοικία του. και μόνο το 5% των πόρων σας ε, αποδίδεται στα άτομα με ειδικέ ανάγκες. Με εκπλήσει, πολύ μικρό το ποσοστό αυτό. Πρέπει να κάνουμε περισσότερο για να τους βοηθήσουμε. Για τους υπόλοιπους πρέπει να βοηθήσουμε την επαγγελματική κατάρτιση, να παρέμβουμε εκεί που δεν υπάρχει ανάπτυξη και απασχόληση, να υπάρξει εκεί ανάπτυξη και απασχόληση, να βγουν από τη φτώχεια εκεί που είναι. Ευχαριστώ και ελπίζω να συνεχίσουμε τη θαυμάσια αυτή τη συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ, εκεί πρόεδρο, στην εισηγήτριά μα. Περνάμε στο επόμενο 6, ειδική έκθεση 11. Να δώσω το λόγο και εδώ στην Ηλιάνα Ιβάνοβα. Σας παρακαλώ, 7-8 λεπτά. Γιατί δυστυχώς έχουμε μεγάλη καθυστέρηση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω όντω να συντομεύσω πάρα πολύ την προβλεπόμενη αυτή παρουσίαση και να τηρήσω το χρόνο αγόρευση που μου δώσατε. Λοιπόν, α περάσουμε κατευθείαν στι διαφάνειε. Το θέμα μα αυτή τη φορά είναι το ερευνητικό σχέδιο του ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού για τη διαχείριση νέα κυκλοφορία, το πρόγραμμα ΣΕΖΑΡ. Και το ζήτημα που τίθεται εδώ πέρα, αν είναι όντω έχει επιφέρει προ τη θέμενη αξία και αν όντω έπρεπε να είχαμε χρηματοδότηση από ευρωπαϊκής πλευράς. Τρεις είναι οι φάσεις, καθορισμός, ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή. Ξέρετε, το 2017 είχαμε καλύψει μέσω ειδική έκθεση ε, τι δύο πρώτε φάσει: καθορισμό και ανάπτυξη. Δεν ασχοληθήκαμε τότε με την υλοποίηση, την εφαρμογή, ενώ η σημερινή μα έκθεση επικεντρώνεται ακριβώ στο στάδιο αυτό, στο στάδιο δηλαδή τη εφαρμογή, τη υλοποίησης από τη συνολική χρηματοδότηση 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ, 2,5 δισεκατομμύρια δίνονται ακριβώς για το στάδιο αυτό της εφαρμογής και της υλοποίησης. Βλέπετε εδώ πέρα ποια είναι τα ερωτήματα, τα ελεγκτικά τα οποία θέσαμε σε σχέση με την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, την αποτελεσματικότητα, τις επιδόσεις του συστήματος διαχείρισης της νέας κυκλοφορίας, τι εντοπίσαμε. Βλέπουμε καταρχάς ότι ε, ο κανονισμός για τον εξυγχρονισμό της διαχείρισης νέας κυκλοφορίας επιφέρει προς τη θέμενη αξία, μόνο ότι υπάρχουν κάποιες αδυναμίες είχαμε έναν συντονισμό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να μετριάσουμε τα κακό κείμενα και να έχουμε καλύτερα ωφέλη όσον αφορά τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες. Ο νέος όμως αυτός κανονισμός παρουσιάζει και κάποιες αδυναμίες. Ιδίω αυτό το οποίο εντοπίσαμε είναι ότι υπάρχουν κάποιες δυσλειτουργίες στα πρώτα στάδια εφαρμογής, κάποια κοινά πιλωτικά προγράμματα δεν ήταν αρκετά συγχρονισμένα και δεν μπορούσαν από κοινού να εφαρμοστούν. Δεύτερη παρατήρηση. Η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν εν γέννη περιττή. Και αυτό έχει να κάνει καταρχάς με το ότι το αρχικό σκεπτικό για τη χρηματοδότηση δεν ακολουθήθηκε στη συνέχεια. Ενώ είδαμε ότι η χρηματοδότηση ουσιαστικά πήγαινε σε συγκεκριμένους παραλήπτες από τις αερομεταφορές, ενώ προβλεπόταν να γίνει κάτι τέτοιο, ενώ το 88% πήγε τελικά σε υπηρεσίες εδάφους. Και είδαμε επίσης ότι οι επενδύσεις αυτές θα μπορούσαν να είχαν γίνει και χωρίς την κοινωνική χρηματοδότηση. Μάλιστα είχαν ξεκινήσει και κάποιες διαδικασίες ανάθεσης προτού εγκριθούν συγκεκριμένα ποσά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχαν τα απαραίτητα ποσά μόνο και μόνο από τα τέλη διαχείριση του ενέργειου χώρου που πληρώνουν οι αεροπορικές μεταφορέ. Είδαμε επίση ότι υπήρχαν κάποιες αδυναμίες στην εφαρμογή του προγράμματος δεν υπήρχε απαραίτητη ιεράρχηση προτεραιοτήτων στην αρχή του προγράμματο. Η ομαδοποίηση των ερευνικών προγραμμάτων δεν βοήθησε όμω τον συντονισμό του και υπήρχε και ένα κίνδυνο συγκρούση συμφερόντων, ο οποίο δεν μετριάστηκε παρκώ. Τέταρτη βασική μα παρατήρηση. Οι βελτιώσεις ε, στην ευρωπαϊκή διαχείριση της ενέργειας κυκλοφορίας δεν έχουν επιδειχθεί επαρκώς ακόμα. Σίγουρα η υλοποίηση βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, θα κρατήσει μέχρι το 2025-2026. Παρόλα αυτά αυξάνονται οι κίνδυνοι καθυστερήσεων και κάποιες συστάσεις που κάνουμε στο πλαίσιο της έκθεσής μας. Καταρχάς, θα πρέπει να βελτιωθεί μια καλύτερη στοχοθέτηση για τα κοινά έργα να καταφέρουμε να ενισχύσουμε την αποδοτικότητα των κοινών έργων, μια καλύτερη αναθεώρηση της χρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχουμε μια καλύτερη παρακολούθηση επίσης όσον αφορά τα πραγματικά ωφέλη από τις επενδύσεις αυτές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε κατά τρόπο οριζόντιο να παρακολουθούμε και να αξιολογούμε καλύτερα τις επιδόσεις του προγράμματος αυτού. Ολοκληρώνω πολύ γρήγορα και προσβλέπω στις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις σας. Να ευχαριστήσω λοιπόν ε, την εισηγήτρια και θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντινόλφη, εισηγητή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Να ευχαριστήσω την κυρία Ιβάνοβα για την εξαιρετική της εργασία Έχω συντάξει, μάλλον έχει συντάξει μια σύντομη έκθεση, το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, η οποία όμω αναφέρεται σε κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα. Καταρχά, προκειμένου να εξηγήσω λίγο καλύτερα τα πράγματα στου συναδέλφου. περί τίνο πρόκειται να κάνω μια γρήγορη περίληψη. Οι αεροπορικέ μεταφορέ είναι πάρα πολύ σημαντικέ γενικότερα για τον ευρωπαϊκό βιομηχανικό τομέα και βέβαια για τι μεταφορέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμβάλλει πάρα πολύ στην κινητικότητα αγαθών υπηρεσιών και πολιτών βέβαια και συμβάλλει πάρα πολύ στην οικονομική ανάπτυξη, τις εμπορικές ανταλλαγές και την απασχόληση. Το 2017 είχαμε περίπου ένα δισεκατομμύριο επιβάτες και 16 εκατομμύρια αγαθά στα αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φτάσαμε σε 11 δισεκατομμύρια πτήσεις το 2017, 30.000 μάλιστα την ημέρα και είδαμε ότι περίπου 37.000 αεροπλάνα σε καθημερινή βάση διασχίζουν τον, ευρωπαϊκό ουρανό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να ρυθμίσουμε την, την κυκλοφορία αυτή την αεροπορική και γι' αυτόν τον λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από το 2000 ξεκίνησε τις απαραίτητες ε, δραστηριότητες με έναν ορίζοντα του 2020. Αυτή τη στιγμή ασχολούμεθα με το τρίτο στάδιο του ΣΕΖΑΡ, δηλαδή με την πραγματική εφαρμογή, υλοποίηση του προγράμματος αυτού στους ευρωπαϊκούς ουρανούς. Αναφερόμαστε εδώ πέρα στο εξής μέχρι να ξεκινήσει το ΣΕΖΑΡ είχαμε μία μεμονωμένη διαχείριση της ενέργειας κυκλοφορίας από κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά. Έρχεται τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το σχέδιο αυτό να ενοποιήσει την διαχείριση της ενέργειας κυκλοφορίας στους ευρωπαϊκούς ουρανούς. Χρειάστηκαν λοιπόν να χρηματοδοτηθούν συγκεκριμένα προγράμματα και μας λέει το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο ότι θα μπορούσε εδώ πέρα να μην είχε γίνει η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Για την περίοδο 2014-2020 είχαμε 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν κατανεμήθηκαν βέβαια ομοιογενώς. Βλέπουμε Κυρία Ντινόλφη, μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο αργά, λέει η Πρόεδρος, γιατί τη χαιρένεται το έργο των διερμηνέων. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά αεροδρόμια τα οποία έχουν αποφεληθεί από το σχέδιο ΣΕΖΑΡ και έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις. Από την άλλη βλέπουμε όμως ότι οι περισσότερες επίγειες υπηρεσίες έπρεπε από μόνες τους να χρηματοδοτήσουν τη λειτουργία τους και ενδεχομένω να ζημιωθούν από την όλη αυτή διαδικασία. Σε ποιο βαθμό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαχειριστεί την υλοποίηση του ΣΕΖΑΡ από το 2011 και μετά και κατά ποιον τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συμβάλει πραγματικά στο να δημιουργηθεί ένα ομοιόμορφο ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Μέσω του ΣΕΖΑΡ προβλέπεται ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο και μια ενιαία χρηματοδότηση. Το έχουμε δει όμω αυτό στην πράξη. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε εδώ πέρα αν υπάρχει μια πραγματικά ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία από το πρόγραμμα ΣΕΖΑΡ και αν τα κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση όντω έχουν οδηγήσει σε μια αύξηση των επιδόσεων για την διαχείριση της Ευρωπαϊκής Ενέργειας Κυκλοφορίας. Το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο έλεγξε αν η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως τα πιλωτικά προγράμματα, όντως ήταν επωφελής για τους δικαιούχους, για τους οποίους ήταν πάρα πολύ σημαντικό να ελοποιηθούν συγκεκριμένα προγράμματα εξυγχρονισμού της διαχείρισης της ενέργειας κυκλοφορίας. Εδώ πέρα το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο μας λέει ότι η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πήγε σε δικαιούχους που δεν χρειάζονταν τη χρηματοδότηση και ουσιαστικά κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργείται, αν θέλετε, ένα αντίκτυπο αδράνεια για κάποιου δικαιούχου οι οποίοι θα μπορούσαν με διαφορετικό τρόπο να είχαν χρηματοδοτήσει τι επενδύσει του. Θεωρήθηκε λοιπόν περιττή η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επιδοτήσεις στην περίπτωση αυτή λοιπόν θεωρήθηκαν αναποτελεσματικές για τον κοινοτικό προϋπολογισμό καθότι όπως σας είπα χρηματοδοτήθησαν επενδύσεις που θα μπορούσαν να είχαν χρηματοδοτηθεί διαφορετικά. Το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο μας λέει ότι συγκεκριμένοι φορείς θα μπορούσαν να είχαν προχωρήσει χρηματοδοτικά με τις επενδύσεις αυτές ακόμα και αν δεν υπήρχε η χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό ήταν εντελώ περιττή ουσιαστικά η ευρωπαϊκή χρηματοδοτική στήριξη. Μα λέει επίση το ελεκτικό συνέδριο ότι όλα αυτά τα έργα τα οποία ελέγχθηκαν από του Ευρωπαίου ελεγκτέ θα μπορούσαν να είχαν συμπεριληφθεί στα εθνικά προγράμματα βελτίωσης της ενέργειας κυκλοφορίας. Αυτό είναι ακόμα πιο σοβαρό. Δηλαδή, συγκεκριμένες οι υπηρεσίες θα είχαν μεταθέσει το κόστος αυτό στους τελικούς χρήστες. Κατά αυτόν τον τρόπο, σε ορισμένε περιπτώσεις έχουμε, αν θέλετε, μια διπλή χρηματοδότηση, η οποία έρχεται αφενός από την Ευρωπαϊκή Ένωση και φετέρου από τους τελικούς χρήστες, οι οποίοι χρηματοδότησαν μέσω τελών και φόρων συγκεκριμένες επενδύσεις. Νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να δούμε ότι υπήρχαν για συγκεκριμένε επενδύσεις πολύ αυξημένα έσοδα. Οι αεροπορικές αυτές υπηρεσίες, όπως σας είπα, είχαν ήδη περάσει στον τελικό χρήστη συγκεκριμένο κόστος, ενώ παράλληλα λάμβαναν και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τα κοινά σχέδια, είδαμε τα περισσότερα δεν ήταν όριμα και δεν απαιτούσαν όλα μία συγχρονισμένη υλοποίηση προκειμένου να έχουμε υψηλότερα επίπεδα επιδόσεων. Επίση, το ελεγκτικό συνέδριο μα λέει ότι υπήρχαν συγκεκριμένε τεχνολογίε, οι οποίε την ώρα τη εξολόγηση δεν ήταν ακόμα όριμε και για τι οποίε θα έπρεπε να είχαν γίνει περαιτέρω προσπάθειε έρευνα και ανάπτυξη, προκειμένου να είναι πραγματικά αποδοτικέ. Απουσία επίση κυρώσεων για τη μη τήρηση των κανόνων και αυτό ζημιώνει τελικά την εφαρμογή του κοινοτικού κανονισμού. Μας λέει το ελεκτικό συνέδριο ότι καμία Εθνική Αρχή Επιτήρηση και Εποπτεία δεν έχει την απαραίτητη χρηματοδότηση προκειμένου να μπορεί να παρακολουθεί αποτελεσματικά και εκ του σύνεγγυ τον τρόπο που λειτουργούν οι εθνικέ υπηρεσίε διαχείριση τη ενάρεια κυκλοφορία. Νομίζω ότι εδώ πέρα θα έπρεπε να γίνει μια ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Απουσία τη ιεράρχηση αυτή, η κοινοτική χρηματοδότηση πάλι πήγε σε ε, προγράμματα τα οποία δεν απαιτούσαν ουσιαστικά τη χρηματοδότηση αυτή, ενώ άλλα την είχαν περισσότερη ανάγκη. Επίσης μας λέει το λεκτικό συνέδριο ότι η ρύθμιση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης τελικά έδωσε μια κάποια προστιθέμενη αξία στο όλο σύστημα τουλάχιστον στα πρώτα στάδια του προγράμματος αυτού. Παρόλα αυτά είδαμε ότι στο στάδιο της εκτέλεσης περιλαμβάνοντας συγκεκριμένε λειτουργίες οι οποίες δεν θα έπρεπε ουσιαστικά να είχαν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωση για τον εξυγχρονισμό της διαχείριση τη νέα κυκλοφορία ήταν εν γέννη περιττή και δεν θα έπρεπε να είχε δοθεί όλο αυτό το ποσό χρηματοδότησης εν κατακλείδη από, τον, από την έκθεση αυτή του ελεγκτικού συνεδρίου, καθώ επίση και μέσω άλλων εκθέσεων που είχαμε στην δική μας την Επιτροπή εμφανίζονται συγκεκριμένε αδυναμίες όσον αφορά τη χρηματοδότηση του ΣΕΖΑΡ. Νομίζω ότι υπάρχουν περισσότερες γκρίζες ζώνες τελικά στο ΣΕΖΑΡ παρά σαφή ξεκάθαρα στοιχεία. Και νομίζω ότι εν τέλει μπορούμε να πούμε ότι έγινε μια κακή χρήση του δημόσιου χρήματος, η οποία είναι ζημιογόνος τελικά για τον κοινοτικό προπολογισμό και γι' αυτό το λόγο η δικιά μου η άποψη είναι σαφώς αρνητική για το πρόγραμμα ΣΕΖΑΡ και σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι θα μπορούσαν τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων να είχαν δαπανηθεί διαφορετικά. Να ευχαριστήσω πάντως την κυρία Ιβάνοβα για την εξαιρετική της έκθεση, την εξαιρετική της εργασία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. So, ε, nun darf ich... Λοιπόν, σειρά έχουν οι σκιώδεις εισηγητές. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Γκραπίνη. Ε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την λεπτομερέστατη παρουσίαση της κατάστασης. Να ευχαριστήσω επίσης και την κυρία Ιβανόβα για ε, την ε, ρεαλιστική παρουσίασή της με τα προβλήματα που έχουν συναντήσει στην ΕΣΕΣΑΡ αλλά και ε, σε τη φορά τους στόχους που έχουν τεθεί. Είναι πράγματι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο το οποίο έχει αυτές συνέπειες στην ε, ασφάλεια της αεριναρίας κυκλοφορίας. Χθε στην Επιτροπή Μεταφορών συζητούσαμε ακριβώς το ίδιο πράγμα και δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να βρούμε έναν ε, τρόπο κοινή ε, διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ουρανού. Έχω κάποιες ερωτήσεις για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να, για να συμπληρώσω και αυτά που είπε ο εισηγητής. οι πόροι από το συνδέοντα στην Ευρώπη. Γιατί χρησιμοποιούνται με κανόνες που επιτρέπουν τη σύγκρουση συμφερόντων, δηλαδή σε περιπτώσεις όπου ορισμένοι δικαιούχοι εξετάζουν, εγκρίνουν ε, οι ίδιοι τις αιτήσει τους. Γιατί συμβαίνει αυτό. Το ελεκτικό συνέδριο λέει ότι υπάρχουν κάποια project τον οποίο η εφαρμογή δεν θα τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα. Έχετε να μας πείτε κάτι σχετικά με τις συστάσεις του ελεκτικού συνεδρίου και τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε έτσι ώστε να μειωθούν αυτοί οι κίνδυνοι καθυστέρησης που εντόπισε το ηλεκτρικό συνέδριο. Να ευχαριστήσω το ηλεκτρικό συνέδριο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ε, απαντήσεις της προκαταβολικά. Ελπίζω να λάβουμε απαντήσεις έτσι ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση, η οποία κάθε άλλο παρά ιδανική είναι. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα και εγώ να ζητήσω το λόγο και να πω ότι αυτή η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου μου δίνει την εντύπωση ότι χρειάζεται μια εξειδικευμένη επιτροπή για να την αναλύσει, διότι Πρόκειται για πολύ συγκεκριμένα εξειδικευμένα ερωτήματα. Τα τελευταία χρόνια ασχολήθηκα πολύ με την εναέρια κυκλοφορία και από την εμπειρία μου μπορώ να πω ότι η κυρία Γκραπίνη έχει απόλυτο δίκιο. Σε πολλούς ε, τομείς έχει αποδειχθεί επιτυχημένο το πρόγραμμα, όμως αυτά που διαβάζω στην έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου είναι ότι υπάρχουν πολλές εθνικές κατευθύνσεις, απόψεις. Και αυτό δυσκολεύει την κατάσταση, διότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πείσουμε τα κράτη να ε, παραχωρήσουν αυτές τις εθνικές αρμοδιότητες και να επιτύχουμε τους στόχους μείωσης του διοξιδίου του άνθρακα, κάτι το οποίο αποτελεί στόχο του εννέου ευρωπαϊκού ουρανού. Επίσης υπάρχει ανάγκη για τεχνική διαλειτουργικότητα, κάτι το οποίο δεν βρήκα στην έκθεση. Υπάρχει τεχνολογία η οποία δεν είναι διαλειτουργική αυτή τη στιγμή και αυτό μας οδηγεί πάλι στην αφετηρία. Υπάρχουν ουσιαστικές ελλείψεις σε πολλούς τομείς. Για παράδειγμα, δεν ξέρουμε αν ένα μεμονωμένο αεροδρόμιο μπορεί να υποστηρίξει συγκεκριμένε ε, τεχνολογίε. Μπορεί να είναι δυνατό να το κάνει. Όμω το σύνολο είναι το ζητούμενο. Εάν το σύνολο δεν μπορεί να στηρίξει του στόχου του νέου ευρωπαϊκού ουρανού, τότε δεν θα γίνει τίποτα. Όντω ε, υπάρχει ανεπάρκεια, υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχει κοντόφθαλμη εθνική προσέγγιση από τα κράτη-μέλη. Εθνική έλεγχοι της εναέριας κυκλοφορίας οι οποίοι ε, δυσχεραίνουν τα πράγματα και δυσχεραίνουν και τον ανταγωνισμό. Ο νέος, λοιπόν ευρωπαϊκό ουρανό ε, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τα εθνικά συστήματα. Τώρα σε ό,τι αφορά τι ε, αποκήρυξεις, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Θα ήθελα όμως να εκφράσω τις αμφιβολίες μου για ορισμένα πράγματα που άκουσα. Ο κύριος ε, Μαρινέσκου, που έχει ασχοληθεί και αυτός πολύ με το θέμα, δεν μπορεί να έρθει σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν και παίρνω εγώ το λόγο για εκείνον. Ακριβώς λοιπόν εξαιτία των προβλημάτων που έχουμε με τα κράτη-μέλη έχουμε αντιμετωπίσει δυσκολίες. Ε, οι δυσκολίες όμως αυτές δεν οφείλονται σε προβλήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό λοιπόν θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει σε αυτά τα σχόλια και τις ερωτήσεις και μετά στο ελεκτικό συνέδριο. Thank Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Ευχαριστώ για την συζήτηση. Εισαγωγικά. Θέλω να επενέσω το ελεγκτικό συνέδριο για την εργασία του. Όπως υπεγράμμισαν και πολλοί από εσάς, Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, άμα δούμε τα πορίσματά της και την ε, αναλυτική ανάλυση, μας βρίσκει σύμφωνος. Δεχθήκαμε όλες τις συστάσεις που παρουσίασε το ελεκτικό συνέδριο. Και τι θα κάνουμε για να εφαρμόσουμε αυτές τις συστάσεις. Γιατί παρακολουθούμε πολύ στενά την εργασία του υπευθύνου ανάπτυξης και την εφαρμογή του πιλωτικού προγράμματος μέσω συναντήσεων, τεχνικών ελέγχων, ε, επιτόπου επισκέψεων Αλλά γνωρίζουμε επίσης και καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να υπάρξει επιτάχυνση. Οπότε είναι πολύ επίκαιρα τα απορίσματα και οι συστάσεις του ελεκτικού συνεδρίου. Θα τις λάβουμε υπόψη. Συντόμως. Πρόκειται για πρωτοπόρο προσέγγιση. Και γι' αυτό θα μπορούσε να έχει κάποιες αδυναμίες που δεν, μπορούσαν, δεν θα μπορούσαν ούτε και συλλογικά να έχουν προβλεφθεί όταν ενεκρίθη ο κανονισμός από τους συνομοθέτες. Και γι' αυτό ο κανονισμός περιέχει και μια ρήτρα αναθεώρησης. Πρέπει λοιπόν να αναθεωρήσουμε τώρα την νομοθεσία για να αντιμετωπίσουμε τα, τις αδυναμίες. Ολοκληρώνουμε την αναθεώρηση του κανονισμού και θα προτείνουμε ένα αναθεωρημένο κείμενο εντός του επομένου 12 μήνου. Ποιες αδυναμίες θα αντιμετωπιστούν από αυτήν την αναθεώρηση και θα αναλυφθούν ή τουλάχιστον εξετάζονται δύο διορθωτικές δράσεις. Ορισμένα ήδη περιλαμβάνονται στις ε, συμβατικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο αρμόδιος για την ανάπτυξη του ΣΕΣΑΡ. Όλα αυτά θα επηρεάσουν τις προτεραιότητες των επενδύσεών μας. Ούτως ώστε να περάσουμε από την πιλωτική φάση στην το, στη φάση του κοινού προγράμματος 1 σύμφωνα πλήρως με, την, με τον κανονισμό και με πλήρη ανάλυση κόστους κόστους-οφέλους. Για να απαντήσω στην ερώτηση της κυρίας Γραπίνη, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και αποδίδουμε ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα αυτό της σύγκρουση συμφερόντων. Δεν έχουμε στοιχεία ότι έχει προκύψει κάτι τέτοιο αλλά επειδή υπάρχει κίνδυνος Ζητήσαμε λοιπόν από τις αρμόδιες αρχές να διορθώσουν αυτή την κατάσταση στις επόμενες ε, προκηρύξεις. Υπάρχει όμως απόλυτη ανάγκη να εφαρμοστούν μόνο τα αναγκαία προγράμματα. Δώστε μου λίγο χρόνο ακόμη, είναι πολύ σημαντικό. Συμφωνούμε απόλυτα με τους στόχους που θέτει το συνέδριο ότι πρέπει να δαπανώνται χρηστά οι πόροι. Θεωρούμε ότι οι μέχρι στιγμής επενδυθέντες πόροι δαπανήθηκαν σωστά, αλλά πρέπει να πούμε ότι πρέπει να γίνουν κάποιες βελτιώσεις. Θα συνεχιστεί η χρηματοδότηση για την ανάπτυξη του ΣΕΣΑΡ, αλλά πρέπει να εστάσουμε καλύτερα στις προτεραιότητές του και να ψάξουμε και άλλους τύπους κινήτρων ή αντικινήτρων για να συμπληρώσουν να, ή να υποκαταστήσουν τις επιδοτήσεις. Όπως κάνουμε και με το ΣΕΦ 2 και την επόμενη φάση λοιπόν του εγχειρήματο αυτού. Πρέπει να εστιάσουμε καλύτερα. Να εστιάσουμε στο συντονισμό, συγχρονισμό και διαλειτουργικότητα όλων των επιμέρους προγραμμάτων. Στην περαιτέρω συζήτηση για το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και τη στήριξη του Κοινοβουλίου. γιατί θα έχουμε δυσκολίες στις συνεννοήσεις με τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Τα προβλήματα με τα κράτη-μέλη μας είναι γνωστά. Το ελεκτικό συνέδριο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας. Όντως, ο κατακαιρματισμός της διαχείρισης ενέργειας κυκλοφορίας είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό ε, χρειάζεται ε, βελτίωση. Υπάρχουν ακόμα κάποια ζητήματα οικονομικής διαχείρισης, όπως αναφέρουν οι σκιώδεις εισηγητές, και ο εφιστάμενος μηχανισμός χρηματοδότησης απαιτεί ορισμένοι δικαιούχοι, να ελέγχουν οι ίδιοι τις ε, εφαρμογές τους, τη δουλειά τους και αυτό πιθανώς αποτελεί σύγκρουση συμφερόντων. Είναι κάτι που δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς. Για το λόγο αυτό έχουμε συστήσει να εστιάσουμε στα κοινά έργα και στα ωφέλη τους και να γίνει αναθεώρηση της ε, οικονομικής στήριξης της διαχείρισης ενέργειας κυκλοφορίας διασφαλίζοντας ταυτόχρονα καλύτερη εποπτεία, καλύτερο έλεγχο. Επίσης, κύριε Πρόεδρε, ρωτήσατε κάτι για τις τεχνικές επιτυχίες και να πω ότι υπάρχουν αναφορές σε αυτό στην έκθεση, για παράδειγμα στην έλλειψη ετοιμότητας, επίσης στην σελίδα 19 της έκθεσης ε, αναφέρουμε συγκεκριμένα τεχνικά παραδείγματα και είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι πάντα προσπαθούμε να πετύχουμε τη σωστή ισορροπία ε, και να καλύπτουμε μεν τεχνικές πτυχές, αλλά να ασχολούμαστε και ε, γενικότερα. Ο σκοπός της ανάλυσης είναι να εντοπίσει το πρόβλημα ε, που μας εμποδίζει στην ενοποίηση του Ευρωπαϊκού Ουρανού και αυτό είναι ο κατακαιρματισμός στην παροχή υπηρεσιών, το οποίο έχει επιπτώσει στις ικανότητες, στην αποδοτικότητα και στην παροχή υπηρεσιών. Επίσης, ασχολούμαστε μέσω των συστάσεων με τεχνη... Ε, πιθανότητες τεχνικής αντιμετώπισης του προβλήματος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ το ελεγκτικό συνέδριο. Ξέρω πολύ καλά πως δεν είναι εύκολη η δουλειά σας. Ιδιαίτερα όταν μας λέτε ότι τα κράτη-μέλη δεν είναι ιδιαίτερα συνεργάσιμα και πρόθυμα. Αυτό σίγουρα περιπλέκει τα πράγματα, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για ένα τόσο δύσκολο project. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ο κύριος συγητής ίσως έχει κάποια καταληκτικά σχόλια ή μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Και ο κύριος Αντινόλφ είναι ικανοποιημένος. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν σε αυτό το σημείο και να ε, τη λήξη της ε, κανονικής συνεδρίασης για να περάσουμε στους συντονιστές. Σας ευχαριστώ πολύ.